Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα περάσουμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με τον Εμβέρα Οτζά, Υπουργό Εξωτερικών του Κωσυφοπεδίου. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά στην Επιτροπή μας εκ μέρους του συναδέλφου Έντουαρ Κούκαν, του Προέδρου της ε, Αντιπροσωπείας για τη σχέση με την Νοτιοανατολική Ευρώπη, να καλωσορίσω τον κύριο Εβέρ Χότζα, Υπουργό Εξωτερικών του Κωσυφοπαιδίου. Κύριε Υπουργέ, οι πολιτικές δραστηριότητες τον τελευταίο καιρό στο Κωσυφοπαίδιο ήταν εντονότατες με πολλά γεγονότα και πολλές δραστηριότητες και μάλιστα μετά μια λαθάρουσα περίοδο εξαιτία των εκλογών η νέα κυβέρνηση άρχισε το έργο της προκειμένου να ανταποκριθεί στις πολυάριθμες προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε. Με ιδιαίτερη χαρά μάθαμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση στα πλαίσια του διαλόγου Βελιγραδίου Πρίστινας τα αποτελέσματα ήταν αίσια και μάλιστα επιτεύχθη συμφωνία για πολύ σημαντικά σημεία όπως είναι η ελεύθερη διακίνηση, η αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων και τίτλων σπουδών και ανακοίνωση πληροφοριών για την κατάσταση των την προσωπική κατάσταση. Χαίρομαι και συγχαίρω και τους, ε, τις δύο πλευρές για τις επιτυχίες αυτές. Περιμένουμε τις ε, πληροφορίες σας για τις δύο αυτές συμφωνίες και την εφαρμογή τους και γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ της ελάφρυνσης των διατυπώσεων για την ε, απόκτηση θεώρησης και θέλουμε αμελητή να ξεκινήσουμε το διάλογο για τις θεωρήσεις με τη χώρα σας. Βέβαια, αυτή η ελάφρυση των διατυπώσεων προϋποθέτει μια πλήρωση κριτηρίων από το κοσυφοπαίδιο σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή και την επανένταξη σε τοπικό επίπεδο ανθρώπων που επαναπατρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε λοιπόν την ενεργό συμμετοχή στο τομέα αυτό και περιμένουμε και τις δικές σας προσδοκίες ό,τι αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων και την πρόοδο στο θέμα αυτό. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο και η συζήτηση θα ακολουθήσει τις ομιλίες σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Members of, uh, Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για την παρουσία μου εδώ σήμερα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία και τη δυνατότητα που μου δίνετε για να σας μιλήσω. Είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτή για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας και μια και ε, ήμουνα περίπου μια οκταετία βουλευτής στη χώρα μου, είμαι ιδιαίτερα πρόθυμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η ομιλία μου καλό θα είναι να είναι σύντομη. Δεν χρειάζεται να σας κουράσω με μακροσκελείς εξηγήσεις για να έχουμε χρόνο για τη συζήτηση. Θα ήθελα καταρχήν να σας ενημερώσω ότι η δημοκρατία του Κωσυφοπεδίου είναι μια νέα χώρα και νομίζω ότι συνέβαλε στην ειρήνη, τη δημοκρατία και τη σταθερότητα στην περιοχή. Θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω ότι την τελευταία τριετία καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα κράτος και μια κοινωνία εκ του μηδενός. Και αυτή η διαμόρφωση και εδραίωση του κράτους έγινε χάρη στην υποστήριξη πολλών χωρών και κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που πραγματικά συνέβαλαν και βοήθησαν τα μάλα το λαό του Κωσυφοπεδίου, ο οποίος και είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για την υποστήριξη αυτή. Όπως επισήμανε και η Πρόεδρος, τους τελευταίους μήνες είχαμε μια συνταγματική κρίση στο Κωσυφοπέδιο. Ε, χρειάστηκε να παραιτηθούν δύο πρόεδροι και ως νεοπαγής χώρα χρειάστηκε να βρούμε μια λύση. Καταφέραμε να βρούμε αυτή τη λύση και τελικά να εκλέξουμε ένα νέο πρόεδρο που είναι και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των Βαλκανίων. Και εκπροσωπεί τη χώρα μας και μάλιστα η πρόεδρος αυτή είναι υπερκομματική, δεν έχει ιδιαίτερη κομματική υποστήριξη, απόχρωση φυσικά είναι υπέρ της, του σεβασμού του κράτους δικαίου, θα υποστηρίξει την εφαρμογή του κράτους δικαίου και ελπίζουμε να συμβάλλει στην πολιτική σταθερότητα που μας είναι τόσο πολύτιμη και απαραίτητη. Και ε, ως υπερκομματική πρόοδος θα εκπροσωπεί το σύνολο της κοσοβάρικης κοινωνίας. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να φέρω είναι τα τελευταία τρία χρόνια. Ο στόχος μας είναι η εθνική συνύπαρξη σε αυτή την πολυεθνική κοινωνία που έχουμε. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα συνήλθα στην Πρίστινα 25 χώρες σε μια ε, διεθνή διάσκεψη και έγινε μια επισκόπηση της κατάστασης και των επιτευγμάτων μας την τελευταία τριετία και θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι την τελευταία τριετία καταφέραμε να εφαρμόσουμε περίπου το 90% του σχεδίου Αχτισάρη. Και σήμερα το Κόσοφο πέδιο είναι μια πολυεθνική κοινωνία με υψηλό επίπεδο ένταξης των μειονοτήτων. Και την τελευταία τριετία επενδύσαμε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουμε πέντε, νέες, ε, πέντε νέους δήμους, κυρίως ε, με υπεροχή της σερβικής μειονότητας και έχουμε στο Κοινοβούλιο 26 βουλευτές από μειονότητες, από διάφορες μειονότητες. Καταφέραμε λοιπόν να διαμορφώσουμε και πολυεθνικούς θεσμούς εκ του μηδενός και σε κεντρικό και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, κατορθώσαμε ως νέα κυβέρνηση να επικεντρωθούμε στην προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας, της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε πρόσφορο έδαφος για οικονομική ανάπτυξη και τη διεξαγωγή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στο δικαστικό σύστημα, αλλά και στη διοίκηση. Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα να αναφέρει η Πρόεδρος στο διάλογο που έχουμε με το Βελιγράδι. Ο διάλογος αυτός Βελιγραδίου-Πρίστινας ξεκίνησε με το ε, ψήφισμα του ΟΗΕ του περσινού Σεπτεμβρίου Πρόκειται για ένα διάλογο που επικεντρώνεται κυρίως σε τεχνικά ζητήματα. Προς το παρόν καταφέραμε να συνάψουμε τρεις συμφωνίες στα πλαίσια του διαλόγου αυτού. Οι συμφωνίες ε, αφορούν τρία κυρίως ζητήματα. Το πρώτο είναι η αμοιβαία αναγνώριση των ε, τίτλων σπουδών, των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών. Το δεύτερο αφορά την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων και το τρίτο πληροφορίες ε, από δημοτολόγια, ληξιαρχία. Πάντως, ε, στη διάρκεια του έτους είμαστε πρόθυμοι και διατεθειμένοι να συνάψουμε και άλλες συμφωνίες με το Βελιγράδι, γιατί μας ενδιαφέρει πρόοδο στο διάλογο αυτό. Από πλευράς μας ε, θα δείξουμε σοβαρότητα, διαλλακτικότητα και ζήλο προκειμένου ο διάλογος αυτός με το Βελιγράδι να στεφθεί με επιτυχία. Ταυτόχρονα Μας ενδιαφέρουν αγαστές σχέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες. Έχουμε θαυμάσει σχέσεις με τη Μακεδονία, με το Μαυροβούνιο, με την Αλβανία. Και μάλιστα οι σχέσεις αυτές δεν είναι μόνο πολιτικές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα έχουν και εμπορικό και οικονομικό χαρακτήρα. Για να μην μακρηγορήσω και να έχουμε χρόνο για τις ερωταπαντήσεις, θα ήθελα να πω ότι τους επόμενους μήνες βράχει και μέσο πρόθεσμα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρεις μείζονες προκλήσεις. Η πρώτη είναι η ένταξη του βορείου τμήματος του Κωσυφοπεδίου γιατί ε, και έχουμε σερβική κυριαρχία εμείς δεν θέλουμε να δημιουργηθεί μια παγωμένη σύγκρουση στο βόρειο Κωσυφοπέδιο σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε απόσχεση, απόσχεση δεν θα να απόσχεση του βόρειου τμήματος του Κωσυφοπεδίου ούτε θέλουμε να προσφύγουμε σε χρήση βίας αποκηρύσουμε οποιαδήποτε χρήση βίας η δεύτερη πρόκληση είναι οικονομικού χαρακτήρα, αφορά την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πριν από λίγους μήνες επεξεργαστήκαμε και προτείναμε ένα πολύ καλό σχέδιο οικονομικής δράσης με τη βοήθεια των κορυφαίων εμπειρογνωμόνων και του Κωσυφοπεδίου και της ευρύτερη περιοχής και δεν θα αφιστούμε προσπαθειών προκειμένου να βελτιώσουμε την, το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών μας. Τρίτη πρόκληση και πολύ σημαντική αφορά την ενταξιακή προοπτική, τη συγκεκριμενοποίηση της ενταξιακής προοπτικής του Κωσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θα ζητούσαμε την υποστήριξή σας, ιδιαίτερα για τον οδικό χάρτη για τις θεωρήσεις. Από, τους, από τα 50 εκατομμύρια των κατοίκων των Βαλκανίων Μόνο τα 2 εκατομμύρια των κοσυφοπεδίων, των κοσοβάρων δεν ε, δικαιούνται να ταξιδεύουν χωρίς θεωρήσεις. Εμείς θα θέλαμε δεν θέλαμε αποφέτωση του χρόνου κατάργηση των θεωρήσεων, απλώς θέλουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δρομολογηθεί ο δικός χάρτης για τις θεωρήσεις, προκειμένου να εκπληρώσουμε τα απαραίτητα κριτήρια και προδιαγραφές. Ήδη έχει γίνει σημαντική προεργασία, έχει προηλιανθεί το έδαφος την τελευταία διετία. Πάντως, αν μέχρι το τέλη του έτους καταφέρουμε να εγκρίνουμε τον, τον οδικό αυτό χάρτη για τις θεωρίες, θα δημιουργηθεί μια νέα όθηση και σίγουρα η κυβέρνησή μας είναι διατεθειμένη να επιτελέσει το έργο της για να υλοποιηθεί αυτό το όνειρο. Μας ενδιαφέρουν ε, συμβατικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κωσυφοπέδι είναι η μόνη χώρα της περιοχής που δεν έχει συμβατικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο θα μεταμορφώσει τις σχέσεις Κωσυφοπεδίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλλει τα μάλλα στην πολυπόθητη οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κυρία Πρόεδρε, το μόνο πρόγραμμα που έχει μια μικρή χώρα σαν τη δική μας είναι ε, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η ευρωπαϊκή προοπτική, η ενταξιακή προοπτική είναι κάτι που θα μας εξασφαλίσει μια προβλεψιμότητα, μια σταθερότητα και ταυτόχρονα το ιδεώδες πλαίσιο για μια χρηστή διακυβέρνηση και για μεταρρυθμίσεις. και οι μικρές χώρες και τα μικρά έθνη έχουν δικαίωμα ύπαρξης και νομίζω ότι όλες οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς μια ευρωπαϊκή προοπτική. Η ευρωπαϊκή προοπτική είναι το παν για μας. Είναι ο μόνος στόχος, το μόνο πρόγραμμα που έχουμε ως νεοσύστατη χώρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά όλους ε, για την θερμή υποστήριξη των τελευταίων χρόνων και να ευχαριστήσω όλους σας για την υποστήριξη και των γειτονικών μας χωρών. Την περασμένη εβδομάδα συμμετείχα σε μία σύνοδο κορυφής στην Κροατία και αυτό που έγινε τελευταία εξαιτία στην Κροατία και η νέα όθηση που δημιουργήθηκε με την ολοκλήρωση των πρωτοεξιακών διαπραγματεύσεων, αυτή την όθηση θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε και εμείς, αυτή την ορμή να την αξιοποιήσουμε για να συγκεκριμενοποιήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική και για το κοσυφοπαίδιο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας μιλήσω εδώ σήμερα και με φυσικά στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες και ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Αρχίζει η συζήτηση. Θα ήθελα να μην υπερβείτε τα τρία λεπτά συνάδελφοι έτσι ώστε να έχουμε το χρόνο που χρειάζεται για την ημερήσια διάσταση διάταξη. Ο κύριος Έντουαρ Κόκαν έχει το λόγο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω εξ ονόματος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από όσο γνωρίζω είναι πρώτη φορά που βρίσκεστε εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας την τρέχουσα κατάσταση στο Κωσυφοπαίδιο και τις μελλοντικές εξελίξεις μπορώ να σας πω ότι ο διακοινοβουλευτικός διάλογος που προωθούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους ε, ομολόγους μας, με τους εταίρους μας από την αντιπροσωπεία του Κωσυφοπεδίου μας οδηγεί σε πολύ καλές επαφές, σε, κοινές, σε κοινά ανακοινοθέντα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι μπορούμε να σταθούμε σε ουσιώδη ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το κοσυχοπαίδιο. Θα ήθελα επίσης να επιβεβαιώσω το σχόλιο της Προέδρου που είπε στην αρχή ότι μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες σας τις φιλοδοξίες, τα φιλόδοξα σχέδια. Αυτό αφορά και την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων που αναφέρατε. Το Κοινοβούλιο πάντα υποστηρίζει την απελευθέρωση αυτή, διότι όπως είπατε πολύ σωστά, διότι από τα 50 εκατομμύρια των Βαλκανίων, μόνο τα 2 εκατομμύρια δυστυχώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το, το καθεστώς, δεν διαθέτουν θεωρήσεις και θα θέλαμε η Κομισιόν να μην χάνει χρόνο και να αρχίσει τη συζήτηση για τον οδικό χάρτη, για το πώς μπορούμε να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι θα σταθούμε στο πλευρό σας. θα ήθελα να υποβάλω μια σκέψη. Βεβαίως η απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι πολύ σημαντική. Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση των κατοίκων του πεδίου σε σχέση με τους άλλους και θα πρέπει η, η κυβέρνηση να επικεντρωθεί στο θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα πλείονα ζητήματα όπως οικονομικές μεταρρυθμίσεις και άλλες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να υλοποιήσετε για να δείξετε ότι πραγματικά προχωρείτε προς την ε, πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Βεβαίως, απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, αλλά θα πρέπει να σταθείτε και σε άλλους τομείς όπου θα πρέπει να επιτελεστεί πρόοδος. Και δύο άλλα σχόλια θα ήθελα να υποβάλω. Άκουσα κύριε Υπουργέ και μπορείτε ίσως να μας το επεξηγήσετε το ΙΠΕΞ έχει προβάλλει, έχει ετοιμάσει μια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε ένα τέτοιο έγγραφο, ιδιαίτερα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε τώρα. Να δούμε δηλαδή πώς έχει αυτή η στρατηγική, πώς ορίζεται, ποιες είναι οι προτεραιότητες σας και ούτω καθεξής. Θα θέλαμε να σχολιάσετε λοιπόν Μιλήσατε για τον διάλογο που προωθείτε, αλλά γνωρίζουμε ότι η αντιπολίτευση στο Πέδιο έχει επικρίνει θέματα διαλόγου και τη στάση σας σε πολλά θέματα. Από όσο γνωρίζω, θα γίνει μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο για τον διάλογο αυτό Άλλοι μιλάνε για έλλειψη διαφάνειας, για το ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται επαρκώς. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς θα αντιμετωπίσετε τα ζητήματα αυτά, τις επικρίσεις αυτές. Ως προς την ε, απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, ε, σας είπα τι σκέφτομαι, δεν είναι το μόνο θέμα σας καλωσορίζω και πάλι και είμαστε και στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε κύριε Κόκαν. Η κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο, που είναι η συγγήτρια για θέματα κωσυφοπεδίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω εξ ονόματο τη ομάδα μου αλλά και του Κοινοβουλίου τον Υπουργό Εξωτερικών του Κουσφοπεδίου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλώ ορίσατε και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μαζί σε αυτό το διάλογο. Ο κύριο Κούκαρ ανέφερε πολλά από τα σημεία που θα ήθελα και εγώ να θέσω και γι' αυτό θα επικεντρωθώ σε άλλα για να μην επαναλάβω τον προαλήσαντα. Θα ήθελα να πω όμω ότι η αντιπροσωπεία μα για την Νοτιοανατολική Ευρώπη πριν από λίγε εβδομάδε μετέβη στο Κωσυφοπαίδιο. Εντάξει, μήνα, πέρασε μήνα και ώρα στο Μάιο ήταν. Πιστώσαμε εκεί ότι είναι πολύ ενεργό το κοινοβούλιο. Και εγώ είμαι βουλευτή, ξέρω, πολλέ φορέ κυβερνήσει δεν θέλουν να είναι τόσο δραστήρια τα κοινοβούλια, ειδικά όταν τι επικρίνουν. Είναι όμω θετικό μήνυμα ε, τη ε, αναπτυσσόμενη δημοκρατία στη χώρα σα και θα ήθελα να ρωτήσω τι λέει το Κοινοβούλιο, πώς γίνεται εκεί η συζήτηση για το διάλογο Πρίστινας Βελιγραδίου που θα λάβει χώρα αύριο. Θα μεταβώ και εγώ την άλλη εβδομάδα στο κοσυποπέδιο και θα μάθω περισσότερα εκεί. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω ή να σχολιάσω αυτά που λέτε. Έχετε μεγάλο δίκιο ε, τονίζοντας ότι είναι πολύ σταθερή η χώρα πλέον στην περιοχή. Ε, φαινόμενα που βλέπουμε στη γειτονική Αλβανία για παράδειγμα ε, μετά τις εκλογές δεν εμφανίζονται στο Κοσμοπέδιο. Μπορεί αμέσως μετά τις εκλογές να υπήρχαν κάποια μικρά προβλήματα. Τώρα όμως είναι σταθερή κατάσταση, ακόμα και αν το ασπιζητού ορισμένοι. Γίνονται πολλές συζητήσεις, αλλά θετικές οι εξελίξεις γενικότερα που διαπιστώσαμε από τις εκλογές ε, του Δεκεμβρίου και εντεύθεν. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής είπατε ότι θα πρέπει πολύ να καταπολεμήσετε ε, το οργανωμένο έγκλημα και την υπόθεση της διαφθοράς. Ε, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τις νομικές πτυχές, για το Κοινοβούλιο, γιατί μία από τις επικρίσεις που ακούμε είναι ότι δεν υπάρχει νόμος για την προστασία των θυμάτων. Πώς θα μιλήσει ο κόσμος για περιπτώσεις διαφθοράς οργανωμένου εγκλήματος. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και ουσιαστική να προστατεύονται οι ε, μάρτυρες. Μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Έχει ε, τεθεί ενισχύ, προβλέπετε, και το όλο θέμα του προπολογισμού. Ο Πρωθυπουργό ε, προεκλογικά έκανε υποσχέσεις για... Πώς να το πω... Ε, ο προπολογισμό εγκρίθηκε, αυξήθηκαν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, έχετε πρόβλημα με το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Πώς, βλέπετε, πώς προβλέπετε τις εξελίξεις στο μέλλον να μην γίνει το δημοσιονομικό τέτοιο πρόβλημα όπως σε άλλες χώρες αυτό τον καιρό στην Ευρώπη. Και τώρα σε ό,τι αφορά το διάλογο κόσμο Παιδίου Σερβίας έχω επίσης την αίσθηση ότι γίνεται κάποια πρόοδο. Είναι πάρα πολύ καλό καν το γεγονό ότι κάθονται στο ίδιο τραπέζι δύο κυβερνήσεις και προσπαθούν να οικοδομήσουν μια εμπιστοσύνη που στο παρελθόν απουσίαζε. Τι κάνει η κυβέρνησή σας για να πείσει την κοινή γνώμη στο Κωσυφοπέδιο ότι αυτό είναι κάτι προ όφελο του Κωσυφοπεδίου, ότι θα βγει ένα αποτέλεσμα δηλαδή. και όχι για να πάρει ε, πλήρες καθεστώς ε, υποψηφίας χώρας η Σερβία. Γιατί εμεί αυτό συζητούμε αυτόν τον καιρό, οι υποστηρικτέ του πεδίου με την Κομισιόν και το Συμβούλιο, ότι να ε, αποκομίσει κάτι το Πελιγράδι, να αποκομίσει και το πεδίο από τι συζητήσει αυτέ. Και ένα τελευταίο. Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο υπερασπίζεται ε, πάρα πολύ το δικαίωμα ε, των ε, πολιτών του Κωσυφοπεδίου στο να ταξιδεύουν. Το ξέρετε, για το τελευταίο διάστημα τι αποφασίσατε για την επαναπροώθηση και επανιστοχή. Αυτά και καλή δύναμη. Ευχαριστώ η Πρόεδρος. Οι συντονιστές, ο κύριος Σαλαφράνκα πρώτος. Σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι να τηρείτε τους χρόνους σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω και να σας υποβάλω τρία ερωτήματα, πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Μας είπατε ότι έχετε πολύ καλές σχέσεις με τις γείτονες χώρες και θα ήθελα κάπως να μιλήσουμε περισσότερο για τη σχέση σας με τη Σερβία. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η πρόοδος που έχει επιτελεστεί για τη σχέση σας με τη Σερβία και ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία εκκρεμούν. Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, τι προτεραιότητες έχετε ως προς τη σχέση σας με τις ΗΠΑ και πώς προωθείτε ο διάλογος, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε. Επίσης, έχετε άτυπες ή επίσημες επαφές με κυβερνήσεις των κρατών μελών που δεν έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του κράτους. Ο κύριος Παντζέρη, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντάχει θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις και να σας υποβάλω και μερικές ερωτήσεις. Δεν αρνούμε ότι έχει γίνει μία σχετική πρόοδος ως προς την κατάσταση στο κοσυφοπέδιο και δεν αμφισβητούμε τη θέλησή σας να ακολουθήσετε μία πιο ε, σωστή πορεία για το κοσυχοπαίδιο και να μην είναι εικονικές οι θέσεις σας. Όμως ε, τι εννοείτε όταν μιλάτε για σταθερότητα. Υπάρχει η ενεργητική και η παθητική σταθερότητα, όπως είπε και η κυρία Λούνατσεκ. Βλέπω ότι δυστυχώς ακολουθείτε τη δεύτερη οδό και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσετε σε ορισμένους στόχους που είχατε ορίσει αρχικά. Μιλώ για οικονομική και κοινωνική, κοινωνική ανάπτυξη, η οποία θα έπρεπε να είναι επαρκής, δηλαδή να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των κατοίκων του Κωσυφοπεδίου. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από πλευράς νομοθετικού έργου ως προς την αυτονομία της δικαιοσύνης. Υπάρχει το θέμα της δικαιοσύνης που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επίσης, θα πρέπει να καταπολεμήσετε τη διαφθορά και την εγκληματικότητα, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγαλύτεροι θύλακες δημοκρατίας. Δεν θα ήθελα να γίνει μία συζήτηση η οποία ήδη προϋπάρχει. Δηλαδή δεν μιλάμε για μία προσέγγιση more for more για το πεδίο. Θέλουμε να μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε αν όμως διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πραγματικές εξελίξεις και βελτιώσεις. Θα ήθελα τη γνώμη σας σε σχέση με την ε, γενική συλλογιστική που επικρατεί σε σχέση με το Πέδιο διότι έχετε πολύ καλές σχέσεις με την Αλβανία και την Μακεδονία, αλλά το πρόβλημα έγκυται στη σχέση σας με τη Σερβία. Αν και φαίνεται ότι η Σερβία δέχεται ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει την οδό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποδεχόμενη και το δικό σας κράτος. Θα πρέπει όμως να επιληθεί το θέμα του βορρά του Κωσυφοπεδίου και να υπάρχουν ε, αγαστές σχέσεις με όλες τις γείτονες χώρες. Ως προς θέμα των θεωρήσεων θα ήθελα να σας πω ότι αντικειμενικά δεχόμαστε αυτή την πορεία έτσι ώστε να έχουν περισσότερες ε, δυνατότητες οι, οι Κωσοβάροι αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με, τις, ε, με την πρόοδο που έχει επιτελεστεί όπως σας έχουμε επανειλημμένα ζητήσει. Ο κύριος Κάτσιν από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ και χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έναν άμεσο ε, διάλογο. Και ως εισηγητής για θέματα Σερβίας θα ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να, έχουμε, να υπάρχουν και εκπρόσωποι της Σερβίας από το Κωσυφοπέδιο μέσα σε αυτό το διάλογο μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου. Αυτό το έχω πει πολλές φορές. Πρόκειται για τη σχέση σας με τη Σερβία και οι μειονότητες πρέπει να εμπεριέχονται, να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο. Ήδη ο πέμπτος γύρος έχει αρχίσει και θα πρέπει να προωθηθεί και στο μέλλον και θα ένα πολύ καλό σημάδι, όχι μόνο για τις ε, διμερείς σας σχέσεις και για την καλύτερη πολιτική ατμόσφαιρα, αλλά θα ήταν και ιδιαίτερα θετικό για ολόκληρη την περιοχή, να συμμετέχουν οι μειονότητες στο διάλογο αυτό. Θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για τα πρόσφατα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου, δηλαδή τη συμφωνία το να μπορεί κανείς να περάσει τα σύνορα της Σερβίας μόνο με ταυτότητα. Εμείς δώσαμε μεγάλη μάχη έτσι ώστε να μπορούμε να μεταβούμε στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μόνο με ταυτότητα. Και εσείς τα καταφέρετε. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν επικρίσεις από την Εθνική Συμμαχία, την Κυβερνόσα Συμμαχία και την Αντιπολίτευση ως προς το θέμα. Θα πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Και επειδή το Κωσυφοπαίδιο είναι ένα νέο ε, κράτος με νέους θεσμούς και μία αντιπολίτευση χωρίς πείρα, θα ήθελα να προωθήσετε περισσότερο το διάλογο με την αντιπολίτευση. Γιατί δεχτήκαμε ε, προσώπους από την αντιπολίτευση. Ο κύριος Κούκαν ήταν παρόν και άλλοι συνάδελφοι και ήταν πολύ δύσκολος αυτός ο διάλογος με τη δική τους αντίληψη για το μέλλον του κοσυφοπεδίου που ήταν διαφορετική και τις δηλώσεις τους για την ε, δημιουργία κρατών στην περιφέρεια με την προκλητική του στάση είδαμε ότι αυτό ήταν ε, αρκετά, αρκετά αρνητικό. Δεν ε, βοηθάει ούτε το Κωσυφοπαίδιο, ούτε τις γειτονές χώρες, ούτε την ευρύτερη περιοχή. Η άπειρη αντιπολίτευση θα πρέπει να ενηλικιωθεί και να είναι και πιο μετριόφρον. Η πλειοψηφία λοιπόν φέρει την ευθύνη να προωθήσει αυτό το διάλογο και να κάνει τις σωστές εκτιμήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντανζόν, που είναι ο πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Υπουργέ, κύριε Εμβέρ Χοντζάι. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που ήρθατε εδώ γιατί γνωρίζω και την προσωπική και την επαγγελματική σας ακυριότητα και νομίζω ότι είναι ένα καλό μήνυμα από την ε, κοσοβάρικη κυβέρνηση ο διορισμός σας στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Έχω τρεις παρατηρήσεις για το διάλογο. Εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ενθαρρύνω για τα πολύ θετικά αποτελέσματα του διαλόγου με το Βελιγράδι και στην αρχή του διαλόγου είδαμε ότι η Πρίστινα έχει κάποιες επιφυλάξεις, ανησυχίες, δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Εγώ θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε με δέσμευση και ζήλο αυτό το διάλογο, γιατί θα είναι ζωτική σημασία και για την περιοχή, αλλά και για την ε, στάση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να γίνει χωρίς ιστεροβουλία αυτός ο διάλογος γιατί οι όροι και οι αρχές του διαλόγου είναι σαφείς και μάλιστα τα πρώτα αποτελέσματα μας υπενθυμίζουν το διακύβευμα. Θα πρέπει να βελτιώσετε το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών σας και των Σέρβων πολιτών του, Κωσοφο, Κωσυφοπεδίου. Αυτό είναι ζωτική σημασία και για την περιοχή. Ο διάλογος δεν αφορά το καθεστώς του Κωσυφοπεδίου, δεν πρόκειται να αμφισβητήσει την αναγνώριση που έχει γίνει ήδη από μερικές χώρες, ούτε θα υποχρεώσει το Βελιγράδι να σας αναγνωρίσει αν η Σερβία δεν θέλει να σας αναγνωρίσει και οι δύο πλευρές, και η Σερβική και η Κωσοβάρικη, θα πρέπει να δεσμευτεί πλήρως, καλόπιστα και χωρίς θεροβουλία, γιατί ο διάλογος είναι πραγματικά θετικός. Δεύτερο σχόλιο για την αποστολή ULEX, που είναι η πιο ε, μεγάλη αποστολή μη στρατιωτικής φύσης ε, που έχει αναπτύξει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι στόχο τη αποστολή αυτή είναι να βοηθήσει το Κωσυφοπέδιο Γιατί πολλά σχόλια ακούσαμε στον τύπο και διαβάσαμε, αλλά και σχόλια τη πολιτική τάξη του Κωσυφοπέδιου που αφισβητούσαν την αμεροληψία τη Γιούλεξ και την αναγκαιότητα τη παρουσία τη και του έργου τη, ιδιαίτερα στο δικαστικό τομέα. Νομίζω ότι είναι κέριο θεμελιώδου σημασία να βοηθήσετε εσεί τη Γιούλεξ, γιατί η Γιούλεξ για να σα βοηθήσει είναι στο κοσυφοπαίδιο, για να γίνει ένα πραγματικά κράτο δικαίου και θα πρέπει και η κοσοβάρικη πολιτική τάξη να στηρίξει τη Γιούλεξ και να ε, μην υποβάλει απαξιωτικά σχόλια ή αρνητικά για τη Γιούλεξ. Ό,τι αφορά το πολιτικό κλίμα του Κωσυφοπεδίου, Σίγουρα η κατάσταση προχωρά, προοδεύεται και μας επιθυμήσατε τις πρόσφατες κρίσεις που αντιμετωπίσατε. Εγώ πιστεύω ότι η κοσοβάρικη πολιτική τάξη θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η ακραία πόλωση είτε εξαιτία της πρόσφατης ε, σύγκρουσης ε, είτε εξαιτία των ε, μικροκομματικών παιχνιδιών μια τέτοια πόλωση είναι πολύ επικίνδυνη και έχετε παραδείγματα από τους γείτονές σας με τους οποίους έχετε εργαστεί συνεργασία. Είδατε ότι η άκρατη αυτή πόλωση οδηγεί σε διέξοδο του δημοκρατικού παιχνιδιού και νομίζω ότι η κυβερνούσα τάξη μπορεί να είναι πολύ πιο διορατική και να ξεφύγει αυτή την υπερβολική πόλωση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει και θα συνεχίσουμε με ένα δεύτερο γύρο. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τις ερωτήσεις, τα σχόλιά σας και τις συμβουλές είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί είμαστε νέος σύστατη χώρα, αλλά και εγώ προσωπικά που διατελώ υπουργό Εξωτερικών ε, της χώρας μου, θέλω και είναι πολύ η συμβολή σας σε πολλά θέματα και πάρα πολύ σημαντική. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Μπορεί να είμαι σύντομος για λόγους χρόνου, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας είναι από τις σημαντικότερες ε, υποθέσεις. Η ε, κυβέρνηση εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για να αναπτύξει ε, ένα νέο οικονομικό σχέδιο για την οικονομική ανάπτυξη. Αν όμως, για να τα πούμε ειλικρινά, η χώρα μας είναι η μόνη χώρα που αποκλείεται από όλους τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, τους περιφερειακούς και τους ευρωπαϊκούς ε, για το εμπόριο και την οικονομία ε, δεν είναι και το καλύτερο περιβάλλον για να αναπτυχθεί κανείς οικονομικά. Προς το παρόν λειτουργούμε ως ένα απομονωμένο νησί στο εσωτερικό της περιφέρειάς μας σε σχέση με την Ευρώπη. Και θα σας παρακαλούσα να μας υποστηρίξετε περισσότερο τη χώρα μας να ε, αναπτύξουμε εμπορικές σχέσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. θα καταλαβαίνετε τι είδους υποστήριξη ζητώ σχετικά με το εμπόριο ε, της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο, η στρατηγική μας για την εξωτερική πολιτική. Το τελευταίο διάστημα, 4-5 μήνες, επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ ε, να καταρτήσουμε ένα έγγραφο για την εξωτερική πολιτική και βασικό στόχος είναι να οικοδομήσουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας απασχολεί και όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' αυτή, αλλά με ορισμένα κράτη-μέλη. Εμείς είμαστε μικρή χώρα. Δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε την πολυτέλεια, να έχουμε εταιρική σχέση με όλες τις χώρες του κόσμου. Προσπαθούμε να εστιάζουμε τις δυνάμεις μας και την προσοχή μας. Επίσης, αυτό το έγγραφο ε, φιλοδοξεί να έχει περισσότερη αναγνώριση. Προς το παρόν, όπως γνωρίζετε, 76 κράτη μας έχουν αναγνωρίσει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μας αναγνωρίσουν και άλλα κράτη ανά τον κόσμο και αυτό θα ήταν θετικό και πολύ χαρμόσυνο νέο τις επόμενες εβδομάδες. Και ένα τελευταίο, ίσως και το πρώτο από αυτό το έγγραφο της εξωτερικής πολιτικής, είναι να καθορίσουμε τη σχέση μας και τη θέση μας στην περιφέρεια. Ποια είναι η θέση μας σε σχέση με τους γείτονές μας και με όλους τους γείτονες έχουμε άριστες σχέσεις. Θα έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας το έγγραφο αυτό, γιατί η εξωτερική πολιτική μιας μικρής χώρας σαν τη δική μας είναι ε, κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητούμε με τους βασικούς πρωταγωνιστές. Πάντως, το σημαντικότερο είναι να έχουμε βράχοι πρόθεσμους στόχους και δραστηριότητες μέσω πρόθεσμους και μακροπρόθεσμους με απότερο στόχο την ένταξη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη και να ε, γίνουμε ένα κράτος πλήρως αναγνωρισμένο. Τρίτη ερώτηση. Έγινε μια ερώτηση και πολλές άλλες για το διάλογο. Κοιτάξτε, θα ήθελα να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Για μας ο διάλογος είναι σημαντικότατος για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Πρίστινα και στο Βελιγράδι. Και ενδιαφέρομαστε πάρα πολύ να εργαζόμαστε καλή την πίστη. Η ε, Πρίστινα θα κάνει ό,τι μπορεί για να έχει φυσιολογικές σχέσεις με το Βελιγράδι και νομίζω αυτά που επιτύχαμε τους τελευταίους μήνες, ε, οι πρώτες συμφωνίες είναι πολύ σημαντικά βήματα. Και θέλουμε πραγματικά να αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό για μας. Ταυτόχρονα όμως ε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν συζητούμε το καθεστώς. Ούτε την κυριαρχία, ούτε την εδαφική ακεραιότητα, ούτε την αλλαγή τη ε, της συνταγματικής τάξης στη χώρα μας. Αλλά ο διάλογος είναι για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών μας, τη ζωή τους, την περιφερειακή συνεργασία, επίσης κρίσιμο, και πώς να προετοιμαστούν και οι δύο χώρες, και η Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο, για την ε, ευρωπαϊκή τους προοπτική και την ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ότι σήμερα δεν έχουμε τρεις συμφωνίες, θα είχαμε έξι συμφωνίες υπογεγραμμένες αν είχε δείξει μεγαλύτερη ευελιξία το Βελιγράδι. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το μεγαλύτερο θέμα είναι η εφαρμογή όλων αυτών. Και σήμερα ήρθα να σας πω ότι θα εφαρμόσουμε εμείς ό,τι συμφωνήσαμε, αλλά να δούμε αν θα το εφαρμόσει και το Βελιγράδι. Αν έχει αυτή την προθυμία για τις τρεις πρώτες συμφωνίες που υπεγράφησαν. Η προστασία των μαρτύρων. με το πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Και τι γίνεται με την νομοθεσία. Πρέπει να σας πω ότι εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για να ολοκληρώσουμε το πρώτο νομοσχέδιο για την προστασία των μαρτύρων. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζετε όλοι σας ότι ε, η Ulex έχει το καλύτερο πρόγραμμα η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καλύτερο πρόγραμμα για την προστασία των θυμάτων. Είναι από τα καλύτερα ε, για την περιφέρεια και καλύτερα από άλλα προγράμματα που έχουν, ε, δεν έχουν άλλες χώρες στον κόσμο. Για τον προϋπολογισμό και την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και τη σχέση μας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είμαστε πάρα πολύ προσιλωμένοι στην προσπάθεια να αναπτύξουμε μια νέα σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μια νέα συμφωνία γιατί αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε τους μισθούς, για να σας ενημερώσω λίγο, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Αν ακούσετε ότι αυξήθηκαν 50% οι μισθοί, ένας καθηγητής γυμνασίου παίρνει κατά μέσο όρο 250 ευρώ. Δηλαδή αν αυξηθεί κατά το ίμιση ο μισθός του καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι καμία τεράστια αλλαγή η δαπάνη. Και διαπιστώσαμε ότι η δημόσια υπάλληλη, η δημόσια διοίκηση δεν είχε κίνητρο να εργαστεί ε, με τους μισθούς αυτούς που είχαν στο παρελθόν. Και πολύ απλούστατα εγκατέλειψαν τη δημόσια διοίκηση. Και ε, αυτό είναι στα πλαίσια της συνολικής αναθεώρησης που κάναμε τα τελευταία τρία χρόνια και των μεταρρυθμίσεων. Ε, πάλι με ρωτήσατε για το διάλογο και πώς επικοινωνούμε με την κοινή γνώμη, πώς ενημερώνεται το κοινοβούλιο, τι κάνει η κοινωνία των πολιτών, ενημερεί ο τύπος, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας κτλ. Σε κάθε συνεδρίαση σε κάθε γύρο του διαλόγου δηλαδή, η κοινή γνώμη, τα μίντια, οι βουλευτές ενημερώθηκαν για την πρόοδο του διαλόγου. Αλλά εντάξει, οι απόψεις των ανθρώπων διήστανται και σε ό,τι αφορά το διάλογο. τα κυβερνώντα κόμματα αλλά και μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν πάρα πολύ αυτό το διάλογο και γνωρίζουν ότι είναι διεθνής υποχρέωσή μας και πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με ε, τη ε, Σερβική Δημοκρατία. Για την επανεισδοχή έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα με ε, την τοπική αυτοδιοίκηση προσκλήθηκαν οι δήμαρχοι να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια με συντονισμό, με κονδύλι μεγάλο από τον προπολογισμό και ξέρουμε ότι πολλοί επέστρεψαν και είναι και πρόθυμοι να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία και είμαι βέβαιος ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε πιο συγκεκριμένη πληροφόρηση. για την επανεισδοχή. Έγινε και μια ερώτηση για τη Σερβία. Ποια θα πρέπει να είναι η σχέση μας με τη Σερβία. Θα πρέπει η Σερβία σιγά σιγά να αρχίζει να αποδέχεται την πραγματικότητα και την ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου. Uh, και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε το παρελθόν εμείς έχουμε κάθε προθυμία, όχι μόνο έχουμε πολύ καλή περιφερειακή συνεργασία και διάλογο, αλλά από την περιφερειακή συνεργασία να περάσουμε στην περιφερειακή συμφιλίωση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ καλές και εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά πραγματικά για να καλλιεργούμε ε, τις καλές μας σχέσεις με τις βασικούς πρωταγωνιστές ε, ε, τα κυριότερα κράτη στον κόσμο. Αν έχουμε ε, ε, άτυπη ή επίσημη σχέση με χώρες που δεν μας έχουν αναγνωρίσει, έχουμε, γιατί ξέρετε ότι η πολιτική σήμερα είναι πάρα πολύ περίπλοκο πεδίο. Από τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μας έχουν αναγνωρίσει, η πιο άκαμπτη συνήθω είναι η κοινή του γνώμη παρά η πολιτική τάξη. Αλλά το σημαντικότερο ερώτημα που μου θέτουν ως Υπουργό Εξωτερικό όταν ταξιδεύω τον κόσμο και η πολιτική και τα μέσα ενημέρωση και άλλοι εκπρόσωποι με ρωτούν Μα γιατί δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, πείσει τα πέντε μέλη της που δεν σας αναγνωρίζουν να κάνουν το ίδιο βήμα. Και πρέπει να σας πω, γιατί πολιτικοί είμαστε, ότι είναι από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις να απαντήσω. Είμαι πραγματικά πολύ μεγάλος υποστηρικτής του ευρωπαϊκού οράματος, ευρωπαϊστής και ξέρω ότι χρειάζεται χρόνο μέχρι οι κυβερνήσεις αυτές να ε, πάρουν την απόφασή τους. Πέρυσι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε μία γνωμοδότηση. Το Διεθνές Δικαστήριο μάλλον. Ε, για το κατά πόσο η, ανεξαρτησία, η ανακήρυξη ανεξαρτησίας μας ήταν σύνομη ή όχι, υπάρχει αυτή η απόφαση και δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε κανένα λόγο καμία ευρωπαϊκή χώρα να μην το αναγνωρίσει. Μια σύντομη τελευταία παρατήρηση. Δεν υπάρχει καμία χώρα στην Ευρώπη που να έχει διοικητικό έλεγχο ε, στην επικράτεια μιας άλλης χώρας. Αυτό που συμβαίνει είναι αντιευρωπαϊκή προσέγγιση και προσπαθώ να σας απευθύνω έκκληση για μεγαλύτερη υποστήριξη κατά πόσο συμμετέχουν οι Σέρβοι του Κωσυφοπεδίου στο διάλογο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε ειδικό απεσταλμένο που καλύπτει ε, το διάλογο. Είναι, η γυναίκα είναι η κυρία Δίτα Ταχή. Είναι πάρα πολύ δραστήρια, πάρα πολύ καλή και είναι ενήμεροι λοιπόν και οι Σέρβοι του Κωσυφοπεδίου συμμετέχουν και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλά ενταγμένοι στη χώρα σε όλη την επικράτεια. Τα όσα συνέβησαν ε, στο Βορρά τα τελευταία 10-15 χρόνια είχε να, είχαν να κάνουν περισσότερο με κάποια απόπειρα να δημιουργηθεί ένα είδος παγωμένης σύραξης ε, από πλευρά Σερβίας. Τελευταία λοιπόν απάντηση τώρα. Ο διάλογος με την αντιπολίτευση Νομίζω ότι ανταλλάσσουμε απόψει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο με την αντιπολίτευση, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά ταυτόχρονα ο διάλογο με την αντιπολίτευση καμιά φορά γίνεται έτσι με μεγάλες δηλώσει, με μεγάλα σχέδια. Η μόνη μας μεγάλη ιδέα είναι η ευρωπαϊκή ιδέα. Εμείς θα εργαστούμε πάρα πολύ σκρέτσι ώστε κάποια μέρα, δεν λέω πότε, κάποια μέρα να είμαστε μέλος αυτού του μεγάλου εγχειρήματος. Είμαστε κατά των μονοεθνικών κρατών στα Βαλκάνια. Είμαστε κατά των αλλαγών συνόρων. Και θέλουμε να είμαστε μια ε, κοινωνία όπως ε, είμαστε στο παρελθόν και συνεχίζουμε. Υπάρχουν τρεις παρεμβάσεις ακόμα. Θα ήθελα να μην υπερβείτε τα δύο λεπτά έτσι ώστε ο Υπουργός να μπορέσει να σας απαντήσει. Ο κύριος Άτκινς ζήτησε το λόγο από τους ε, ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με το θέμα της Σερβίας. Νομίζω ότι ο Υφυπουργό Εξωτερικών ή ο Αντιπρόεδρος της ήταν υπέρ της Ευρώπης, μίλησε με καλά λόγια, μίλησε θερμά για το τι πρέπει να γίνει. Αλλά είχα την εντύπωση ότι δεν επρόκειτο παρά για λόγια και θα ήθελα να ασκήσω πίεση, να σας ρωτήσω τι ακριβώς κάνετε με τη Σερβία γιατί είχα την εντύπωση, μάλλον μου ερχόταν ο απόϊχος των Ελλήνων και των Τούρκων, δηλαδή πολλά λόγια και λίγες πράξεις. Μπορείτε να μου το αντικρούσετε. Ο κύριος Μπέλτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ, ειλικρινά. Ε, στη δεκαετία του 90 είχα μεγάλη δραστηριότητα στην περιοχή σας και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω πάει και έχω συζητήσει με νέους επιχειρηματίες και ανησυχώ για το επιχειρηματικό κλίμα στο Κωσυφοπαίδιο. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε γι' αυτό. Και δύο σύντομες ερωτήσεις. Τι ρόλο παίζει η διασπορά του ε, Κωσόβου που είναι πολυάριθμη ανά την Ιφίλιο ε, πώς σας βοηθούν για την οικοδόμηση του κράτου, Ξέρω μερικού που είναι επιχειρηματίε, έχουν πολλέ καλέ ιδέε. Και τελευταία ερώτηση, τι γίνεται με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και για τη σταθερότητα. Τα είπε και ο Άτκιν ε, για την ελευθερία των α, θεωρήσεων. Χρειάζεστε να έχετε ένα πολύ γερό δημοτολόγιο, να ξέρετε ποιοι είναι οι πολίτες σας, τι γίνεται σε αυτή την προσπάθεια. Μπορείτε να μου απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω σκιώδη ηγητή από το Λαϊκό Κόμμα για το Κωσυφοπαίδιο, θα ήθελα και πάλι να υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο όμως με μεγάλη πλειοψηφία έχει απευθυνθεί στις πέντε χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο και απευθύνει έκκληση να το αναγνωρίσουν. Το επαναλαμβάνω σήμερα αυτό, όχι μόνο επειδή είναι σημαντικό για το κοσμοπέδιο, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Θα πρέπει να είμαστε συμπαγείς και συντεταγμένοι σε αυτό το σημαντικό τομέα της πολιτικής. Συγχαρητήρια για την ανάπτυξη της δημοκρατίας στη χώρα σας, συγχαρητήρια για τη βελτίωση των σχέσεών σας με τους γείτονες και δεν ε, θεωρώ ότι η σημασία έχει μόνο η Σερβία. Ξέρουμε ότι ήταν δύσκολο και με άλλε γειτονικέ χώρε. Γι' αυτό καλωσορίζω ακόμα περισσότερο τι καλέ σχέσει σχέσει Μακεδονία, Αλβανία, Μαύροβουνίου και ε, την ιδέα για μια ε, κοινή προσπάθεια και ένταξη με τις χώρες Βίσεγκρατ. Έχω και εγώ ερωτήσεις. Πρώτον, ο συνάδελφο Κατσίνου ρώτησε για τι μειονότητε. Μειονότητε υπάρχουν και στη Σερβία. Στο Πρέσεβο, α πούμε, οι Αλβανοί. Τι γίνεται, έτσι ώστε κατέρωθεν των συνόρων οι μειονότητε να έχουν το ίδιο καθεστώ. Το Σύνταγμα του Κωσυφοπεδίου ε, είναι το πιο προχωρημένο σύνταγμα από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Τι ισχύει όμω για τι μειονότητε στη Σερβία. Η προστασία των μειονοτήτων δεν θα πρέπει να είναι διμερή, εν πάση περιπτώσει αμοιβαία και από τι δύο πλευρέ των συνόρων να είναι το ίδιο επίπεδο, αν θέλουμε να επικρατεί σταθερότητα. Δεύτερον, Είστε ικανοποιημένοι και πώς με την ε, δράση της Γιούλεξ ε, στο Βόρειο Κόσοβο και τη Μητροβίτσα ε, Ένεχετε εκεί, μετέχει πλήρως ή υπάρχουν ακόμα προβλήματα και ποια είναι αυτά. Και μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με αυτά. Χαίρομαι που τα πράγματα αναπτύσσονται τόσο καλά και εξελίσσονται στο 5 αλλά τώρα θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσει, μάλλον η Σερβία θέλει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέω έτσι, πώς μπορεί να εμποδιστεί ε, το να μπλοκάρει κάποιος άλλος τη σχέση Κωσόβου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή κάποιος να ε, καταχραστεί τη θέση του για να οδηγήσει σε εμπλοκή τη σχεση ε, Κωσόβου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχετε σκεφτεί αυτό, το συζητάτε στο διάλογο. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό για να απαντήσει και στου συναδέλφου και να κλείσει. Uh, thank uh, ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση όσον αφορά τις ε, σχέσεις μας με τη Σερβία. Νομίζω θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε μία μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ 2005-2007. Οι διαβουλεύσεις της Βιέννης. Συμμετείχα σε αυτό το διάλογο για τρία χρόνια. Ήταν ε, μία διαδικασία υπό την αγίδα του Μάρτι Αχτισάρη που ήταν ο ειδικό απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών και είχε συγκεκριμένη εντολή μία πρόταση για μία εποπτευόμενη ανεξαρτησία για το κοσυφοπέδιο. Σε αυτή την ε, διαπραγματευτική διαδικασία δεχτήκαμε όλα όσα έπρεπε να δεχτούμε και θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι κατά το 2005, 2007 όταν συμμετείχα σε αυτές τις ε, διαβουλεύσεις ε, δουλεύαμε πολύ σκληρά για κάθε παράγραφο του προγράμματος Αχτισάρη, του σχεδίου Αχτισάρη και σκέφτηκα ότι το 2015 θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο Αχτισάρη, το οποίο κάναμε κατά περισσότερο από 90%. Σήμερα ήδη έχει εφαρμοστεί πάνω από το 90% του σχεδίου Αχτισάρη και νομίζω ότι άλλες διεθνείς ε, συμφωνίες έχουν προωθηθεί και σε άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά αν συγκρίνουμε το τι κάναμε εμείς και το τι έχει γίνει αλλού τα τελευταία χρόνια, τρία χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πολύ περήφανοι για την ε, συμπερίληψη, τη συμμετοχή των ε, μειονοτήτων στα εθνικά δρόμενα. Και αυτό που σας είπα σήμερα δεν είναι μια ωραία, μια όμορφη ιστορία. Ε, δεν σας απήγγειλα ένα ωραίο ποίημα για το τι συμβαίνει. Η Σερβία θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται, να αποδέχεται πια την ανεξαρτησία του κοσυφοπεδίου. Εμείς δεν ελέγχουμε τη ζωή του Βελιγραδίου και το Βελιγράδι δεν μπορεί να μας ελέγχει εμάς. Τη Δευτέρα θα προσέλθει κάποιος από το Βελιγράδι με μία πρόταση και ε, νομίζω τη δεύτερη μέρα, τη Δευτέρα γίνεται αυτό, την Τρίτη ε, γίνεται μια συζήτηση για ε, καταμερισμό ή επιμερισμό ε, αρμοδιοτήτων, για διαχωρισμό κρατών. Μα πού βρισκόμαστε στο 99. Παλινοδούμε. Ίσως οι Σλοβαίνοι φίλοι να συμφωνήσουν μαζί μου. Εμείς ε, ήμασταν ε, μέρος ενός έθνους όπως ήταν και η Σλοβενία κάποτε και η Κροατία. Αυτό αφορά και το Μαυροβούνιο, το οποίο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του το 2006. Εμείς το κάναμε το 2008. Τι κάναμε με αυτό τον τρόπο. Χάσαμε 20 χρόνια και δεν θέλουμε να χάσουμε άλλα 10 ή 20 προβάλλοντας μία ιστοριούλα, μία ιστορία για τα Βαλκάνια όπως ίσχυε το 1999. Προς, προς τη διασπορά μας εκτείνεται από τη Σουηδία, την Ορβηγία μέχρι τη Νότιο Αφρική και από την Πορτογαλία μέχρι τη Νέα Υόρκη. Πολλοί γύρισαν στην πατρίδα τους και έκαναν και πολλές επενδύσεις. Τα τελευταία τρία χρόνια εργαζόμαστε για να χτίσουμε μία κοινωνία και μία οικονομία εκ του μηδενός. Μεταξύ 1999 και 2008 μας ενδιέφερε η ειρήνευση της περιοχής. Τα τρία τελευταία χρόνια κάναμε ό,τι μπορούσαμε και έχουμε δημιουργήσει και ένα Υπουργείο μόνο για τη Διασπορά εδώ και δύο μήνες όπου καλεί όλα τα στοιχεία της Διασποράς να επανέλθουν στην πατρίδα τους. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχολεί και ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα του δημοτολογίου, να έχουμε ένα πλήρες δημοτολόγιο για όλους τους κατοίκους. Ως προς την αλβανική μειονότητα στη Σερβία, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι περισσότεροι ζουν στα σπίτια τους, δεν έχουν ενταχθεί καλά, το, το, η εκπαίδευση δεν είναι η καλύτερη δυνατή και Η σερβική κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την ε, πλήρη ε, συμμετοχή τους και ένταξή τους στον ε, ιστό της χώρας. Και έχουμε και την κατάσταση των Σέρβων στο, στο βορρά και στο νότο. Υπάρχει, υπάρχουν επικρίσεις ε, προς τη Γιούλεξ εξαιτίας της κατάστασης του Βορρά. Και η Γιούλεξ θα πρέπει να είναι περισσότερο δραστήρια σε σχέση με το παρελθόν, ιδιαίτερα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στο Βορρά. Στο Βορρά χρειαζόμαστε ασφάλεια και επικράτηση του, του δικαίου Πρόκειται για μία αποστολή που την χάνει υποστήριξη, μιλώ για τη Γιούλεξ, και σε γενικές γραμμές θα καταφέρνει αρκετά καλά. Ως προς το διάλογο και τις σχέσεις μεταξύ Κωσυφοπεδίου, Σερβίας και Ευρωπαϊκής Προοπτικής. Θα ήθελα να πω ότι και οι δύο χώρες θα πρέπει να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο την ίδια ημέρα αλλά και την ίδια ώρα ενδεχομένως. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που ήταν άκρος ενδιαφέρουσα. Προτείνω στους συναδέλφους να κάνουμε μία μικρή διακοπή πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ. Σειρά μου τώρα να σας ε, καλωσορίσω, να σας ευχηθώ καλημέρα και να περάσουμε στο επόμενο σημείο που προβλέπει μια, δημο... μια με... από κοινού με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη συνεργασία με την Αντιπροσωπεία με τις σχέσεις... Ε, για τη σχέση με τη Λευκορωσία μετά την κατάσταση στη Λευκορωσία και τις προεδρικέ 19 Δεκεμβρίου του 2010. Ε, παραλαμβάνω, η ακρόαση αυτή γίνεται από κοινού με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ω εκ τούτου θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αντζέι Γκζιπ που θα συμπροεδρεύσει σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τη Λευκορωσία και να καλωσορίσω και τον Γιάτσεκ Προτασέβιτς που είναι και ο πρόεδρος αυτής της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στη Λευκορωσία, παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τα συμβάντα. Βέβαια εγκρίθηκαν κάποιε κυρώσει. και ελπίζω η παρουσίαση που θα γίνει από τους προσκεκλημένους να μας κατατοπίσουν καλύτερα για την κατάσταση στη Λευκορωσία. Κύριε Γκζίμπ, έχετε το λόγο. Μουτσουμές, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους συμμετέχοντες σε αυτή την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να παρακολουθούμε εκ του τα συμβάντα στη Λευκορωσία μετά τις προεδρικές εκλογές και τις ε, διάφορες ενέργειες καταστολής και καταπίεσης ε, εις βάρος ε, πρώην υποψηφίων προέδρων αλλά και μέλων της κοινωνίας. Συνεχίζονται δυστυχώς αυτά τα επεισόδια. Ελπίζαμε ότι θα σταματούσαν αυτά τα κύματα καταστολής αλλά δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι συνεχίζονται αυτά τα φαινόμενα καταστρατήγησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίασης της ελευθεροτυπίας και της ε, ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και γενικώ μια ζωφερή κατάσταση στη Λευκορωσία. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους εμπειρογνώμονες μας που συμμετέχουν σε αυτή την ε, κοινή συνεδρίαση. Είναι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες. Ο πρώτος είναι ο κύριος Τζέρμαν, ο ειδικό ε, εισηγητής της Επιτροπής ε, Διεθνού, Διεθνού Ελέγχου και επικεφαλής ε, του επιτελείου της ΟΑΣΕ για την ελευθερία του συναθρίζεστε. Η σχετική απόφαση, η σχετική γνωμοδότηση έγινε από την Ειδική Επιτροπή για τον Έλεγχο της Κατάστασης στη Λευκορωσία και ε, με τη συνεργασία του Διεθνούς Δικτύου ε, για τις οργανώσεις των πολιτών. Ε, θα πρέπει να γίνει μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του συναθρίζεστε. Είχαμε πολλά επεισόδια στις 19 Δεκεμβρίου του 2010 στο Μίνσκ με καταστολή διαδηλώσεων και γενικώ πολλά ανησυχητικά επεισόδια. Ο δεύτερο ε, προσκεκλημένο είναι ο κύριο Εμμανουέλ Ντεκό, που είναι ανεξάρτητο ε, εισηγητή ε, του μηχανισμού της Μόσχας που διορίστηκε τον Απρίλιο από 14 χώρες που συμμετέχουν στο μηχανισμό αυτό της ΟΑΣΕ και μετά τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές του 2010 υπέβαλε μια έκθεση εκ μέρους του ΑΣΕ. Επίσης έχουμε, ε, είναι και καθηγητής ε, στη Σορβόνη, διευθυντής ε, ενός κέντρου ερευνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μελετά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το πρίσμα του δικαίου στα πλαίσια της ΟΑΣΕ αλλά και διεθνείς προδιαγραφές σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία. Τρίτος προσκεκλημένος είναι ο κύριος Αλεξάνδρε Μπιαλιάτσκι, που είναι πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βιάσνα. Η Βιάσνα είναι από τους πιο ενεργούς ακτιβιστές και υπερμάχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία ξεκίνησαν διάφορες διαδηλώσεις ε, και δράσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόθεση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών αλλαγών, αλλά και πολιτιστικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Και το Λευκορωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, πολλές φορές ε, απέτυχε την την καταχώρηση αυτής της οργάνωσης. Χαιρόμαστε που ο κύριος Μπιαλιάτσκι ήρθε στην συνεδρίαση αυτή το δικαστήριο του Μίνσκ δυστυχώς επιβεβαίωσε την αρνητική απόφαση κατά της Βιάσνα που αναγνωρίστηκε ως μη καταγραμμένη οργάνωση οπότε με βάση τον ποινικό κώδικα του, της Λευκορωσίας απειλείται εις βάρος τους ποινή από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια. Δεν δεν ήταν λοιπόν βέβαιο ότι θα μπορούσε να έρθει ο κ. για να, να έρθει να μας παρουσιάσει την κατάσταση για την παρούσα κατάσταση στη Λευκορωσία. Χαιρόμαστε όμως που τελικά έχει αυτή τη δυνατότητα γιατί περιμένω αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα και οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Αυτές είναι οι σημαντικότερες πληροφορίες ό,τι αφορά τα διάφορα στοιχεία αυτής της ε, κοινή συνεδρίασης με συμμετοχή της Υποεπιτρέπης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αντιπροσωπείας για τη σχέση με τη Λευκορωσία και θα ήθελα να προχωρήσουμε τώρα στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκζίπ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Νίλι Τζάρμαν. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε να ε, συνεισφέρω και εγώ στη συζήτηση ως προς την κατάσταση που επικρατεί στη Λευκορωσία. Η εργασία μου εστιάζεται στα γεγονότα της 19ης Δεκεμβρίου 2010, δηλαδή τις διαμαρτυρίες μετά από τις προεδρικές εκλογές και τις διαδηλώσεις. Προσπάθησα να καλύψω τα γεγονότα λεπτομεριακά και θα ήθελα να αναφερθώ στα κύρια γεγονότα εκείνες τις ημέρες και να τα εντάξω σε σχέση με το ε, δίκαιο την εσωτερική ένομη τάξη ως προς το δικαίωμα του συνέρχεστε και την ελευθερία λόγου και τύπου. Όπως ξέρετε, ε, δεν έχει προσχωρήσει η Λευκορωσία στην, ε, ε, στο χάρτη θεμελιωτών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, αλλά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπων, με συγχωρείτε, αλλά έχει προσχωρήσει σε, ε, άλλες, σε άλλους διεθνείς χάρτες και διεθνείς οργανισμούς ως προς συμβάσεις που είναι παρόμοιοι και γι' αυτό θα έπρεπε να δέχονται το δικαίωμα την ελευθερία του συνέρχεστε. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ στα γεγονότα της 19ης ε, Δεκεμβρίου του 2010 και θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με τον νόμο της Λευκορωσίας οι, συγκεντρώσεις αυτές ε, θεωρήθηκαν παράνομες διότι δεν είχαν προηγουμένως ε, κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση. Όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε αποφανθεί και είχε τονίσει ότι τη στιγμή που πρόκειται για μια ειρηνική συγκέντρωση, είτε είναι παράνομη είτε νόμιμη, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το δικαίωμα του συνέρχεστε τη στιγμή που πρόκειται για μια ειρηνική διαδήλωση, δεν θα πρέπει να απαγορεύεται. Οι αρχές λοιπόν είχαν την υποχρέωση να προστατεύσουν αυτό το δικαίωμα του, συνέχε, του συνέρχεστε. Και φάνηκε ότι το απόγευμα προς το βράδυ τήρησαν αυτό το, δέχτηκαν αυτή την ε, συγκέντρωση οι αρχές. Οι αστυνομικές αρχές ε, ήταν παρούσες αλλά δεν έδρασαν άμεσα. Όμως ε, στην αρχή της διαδήλωσης καθώς και στα τελευταία στάδια της ε, διαδήλωσης προς το βράδυ δυστυχώς έγιναν επιθέσεις από τις κρατικές ε, δυνάμεις κατά του Βλαντιμίρ Νικλεεφ ε, που ήταν υποψήφιος και κατά δημοσιογράφων που τον συνόδευαν. Δυστυχώς ήταν δυσανάλογη αυτή η επίθεση και απετέλεσε προηγούμενο για τα ξεσπάσματα που έγιναν αργότερα το βράδυ. Στο κέντρο του Μίνσκ όμως οι διαδηλώσεις ήταν, η διαδήλωση ήταν ειρηνική. Συγκεντρώθηκαν 30.000 άνθρωποι για να ακούσουν τις ομιλίες υποψηφίων προέδρων. Και φαίνεται ότι επικράτησε γενικά καλό ε, κλίμα. Στις 10 παρατέταρτο όμως μερικά στοιχεία άρχισαν να επιτίθενται κατά ενός ε, κρατικού ε, κτηρίου και δυστυχώς δεν υπήρξε καμία πρόκληση για, αυτής, ε, για αυτό το ξέσπασμα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο δηλαδή υπήρξαν στοιχεία που προκάλεσαν αυτά τα γεγονότα που προκάλεσαν δηλαδή προβοκάτορες καθαρά. Τη στιγμή λοιπόν που άρχισε ε, αυτή η επίθεση, δυστυχώς η συγκέντρωση δεν ήταν πια ε, ειρηνική και δεν υπήρξε προστασία. Δυστυχώς βεβαίως δεν υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις ε, γύρω από αυτό το κτίριο και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτά τα στοιχεία χρησιμοποίησαν, το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία για την επίθεση. Χρειάστηκε πολύς χρόνος πριν παρέμβει η αστυνομία, αλλά όταν παρενέβη ήταν πολύ επιθετική, χρησιμοποίησε όπλα για να διαλύσει το πλήθος. Φαίνεται ότι δεν έγινε καμία διάκριση για το ποιος ήταν παρόν και ποιοι ήταν οι στόχοι. Μετά λοιπόν από την επίθεση αυτή η κατάσταση παρέμεινε υπό έλεγχο και δεν υπήρχε λόγος να διαλύσει το πλήθος. Η αστυνομία το έκανε όμως μετά από 30 λεπτά. Δηλαδή καταφέρθηκε κατά του υπολείπου πλήθους και προσπάθησε να διαλύσει τον κόσμο και να προβεί σε προσαγωγές πολλοί προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, δεν προπυλάκησαν την αστυνομία, δεν αντιστάθηκαν, οπότε δεν υπήρχε και λόγος να προσαχθούν. Η κρατική μηχανή θεώρησε ότι αυτή η επίθεση κατά του δημοσίου αυτού κτηρίου δικαιολογούσε την επίθεση της αστυνομίας. Εμείς θεωρήσαμε ότι υπήρχαν διαφορές, δηλαδή ένα μόνο μέρος επιτέθηκε κατά του κτηρίου και δεν είχε καμία σχέση με το υπόλοιπο ε, συγκεντρωθέν πλήθος. Το ΕΔΑΔ θεώρησε ότι μόνο αυτοί που επιτέθησαν κατά του κτηρίου είναι υπεύθυνοι, οι οργανωτές της συγκέντρωσης δεν είναι υπεύθυνοι κατά αυτών των ε, επιθετικών πράξεων. Οι αρχές της Λευκορωσίας έλαβαν διαφορετική θέση και στην ουσία προσήχθησαν και υποψήφοι στις προεδρικές εκλογές που δεν είχαν καμία σχέση με τα βία αυτά γεγονότα. και τις μαζικές επιθέσεις. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση σαν να πρόκειται για δύο διαφορετικά γεγονότα. Δηλαδή, δεν πρόκειται για παράνομη συγκέντρωση και αυτοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τα βία γεγονότα δεν πρέπει να προσαχθούν και να τους απαγγελθούν κατηγορίες οι αρχές της Λευκορωσίας δεν προέβησαν σε μία εμπεριστατωμένη έρευνα σε σχέση με τη βία που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικές αρχές. Ε, υπήρξαν πενιχρά στοιχεία στο κατηγορητήριο αυτών που προσήχθησαν και γι' αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί η κατάσταση γιατί στην ουσία η καταδίκη ήταν εντελώς λανθασμένη και βασίστηκε σε πενιχρά στοιχεία. Ο καθηγητής Δεκό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, ε σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση αυτή να μιλήσω συζητητής της ΟΑΣΕ για τη Λευκορωσία και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή ε, να συμμετέχω σε αυτό το πάνελ με τους δύο κορυφαίους συναδέλφους που επιτελούν αξιολογότατο έργο. Η αποστολή που ανέλαβα στα πλαίσια του μηχανισμού της Μόσχας για την ανθρώπινη διάσταση με πρωτοβουλία 14 χωρών συμμετεχόντων ολοκληρώθηκε τυπικά με την επίσημη παρουσίαση της έκθεσής μου ενώπιον του μόνιμου Συμβουλίου της ΟΑΣΕ στη Βιέννη στις 15 Ιουνίου του 2011. Στην συζήτηση αυτή η τσεχική δημοκρατία εκ μέρους των 14 όπως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και, τα, ε, και οι Ηνωμένε Πολιτείε υιοθέτησαν μια στεναρή και προσεκτική θέση. Ενώ η Ρωσία έδειξε μια διπλωματική τραχύτητα και τυπικά και ουσιαστικά ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ρωσίας είναι ιδιαίτερα προσεκτικά ως προς την κατάσταση της Λευκορωσίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύθηκε πάρα αυτά και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΟΣΕ στα αγγλικά και ελπίζω ότι σύντομα θα είναι έτοιμη και η ρωσική μετάφραση. Ε, τώρα αναπόκειται στα κράτη που συμμετέχουν αλλά και στις, ε, στους θεσμούς της ΟΑΣΕ να εξασφαλίσουν μια συνέχεια αυτής της ε, έκθεσης. Αλλά θα είναι αδύνατο να γυρίσουμε τις σελίδες σαν να μην, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα μετά τις 19 Δεκεμβρίου. Φυσικά η διεθνής επικαιρότητα στρέφει την προσοχή μας σε άλλες κρίσεις, στις όχθες Μεσογείου κυρίως, αλλά δεν θα πρέπει η Αραβική Άνοιξη να καταλήξει σε έναν Ευρωπαϊκό χειμώνα. Σε μια συνέντευξη στη Washington Post τον περασμένο Μάρτιο, ο Λευκορός πρόεδρος έκανε ήδη κάποιους παραλυσμούς με τα επεισόδια στην πλατεία Ταχύρ. Μιλά για πέμπτη φάλαγγα για να καταγγείλει τα κινήματα διαμαρτυρίας που κλονίζουν μέλα τη χώρα. Δύο φωνές υψώθηκαν πρόσφατα εκ μέρους του ΟΑΣΕ για το θέμα αυτό. Πρώτα η κυρία Μιγιάτοβιτς, εκπρόσωπος ε, της ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που την 1η Ιουλίου αποτάνθηκε στον πρόεδρο Λουκασέγκο ζητώντα του να σταματήσει την καταστολή ει βάρο των δημοσιογράφων. Πιο πρόσφατα, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Λιθουανία, ο κύριο Αζούμπαλη, που ασκεί αυτή τη στιγμή την εκπεριτροπή Προεδρία τη ΟΑΣΕ, δημοσίευσε ανακοινοθέν με ημερομηνία 5 Ιουλίου για να αποδοκιμάσει την άσκηση βία ει βάρο φιλελληνικών πολιτών. Πέραν αυτών των δύο επίσημων θέσεων, η σιωπή του ΟΝΤΙΡ, του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι δυστυχώς λυπηρή, όπως και η κατάργηση του σημείου επαφή για τους υπέρμαχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχε έδρα στη Βασοβία. Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο λοιπόν συστήθηκε ο μηχανισμός της Μόσχας, χάρη σε πολλές άμεσες και έμεσες επαφές ε, και με διπλωματικές πηγές αλλά και με την κοινωνία των πολιτών έλαβα γνώση πολλών έγκυρων πληροφοριών και μαρτυριών. Είδα ταινίε, φωτογραφίε και διάφορα ε, σχέδια και πληροφορίε για τα επεισόδια τη 19η Δεκεμβρίου, παρόλο που όλα αυτά δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση για προφανεί λόγου εμπιστευτικότητα. Θα πρέπει να επιθυμήσουμε τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφο 2 του εγγράφου τη Μόσχα, που, προβλέπει, που ε, προβλέπει ότι τα συμμετέχοντα κράτη δεν θα λάβουν κανένα μέτρο ει βάρο προσώπων, οργανισμών ή θεσμών εξαιτία επαφών με την αποστολή εμπειρογνωμόνων ή λόγω κοινοποίηση πληροφοριών σε σχέση με το δημόσιο τομέα. Βέβαια, αυτή είναι μια πολύ σημαντική ανησυχία που έχω αυτή τη στιγμή. Η έκθεση καλύπτει μια περίοδο μερικών μηνών και καθημερινά έχουμε εξελίξεις επιβαρύνοντας τον κατάλογο συστηματικών και κατάφορων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια, σε αυτό το στάδιο μόνο αυστηρά συμπεράσματα μπορούμε να αντιλήσουμε και φαίνεται ότι τα επεισόδια κάποιων ταραξιών άγνωση ταυτότητα μέχρι στιγμή χρησιμοποιήθηκαν ω πρόσχημα για τη βίαιη διάλυση μια ειρηνική διαδήλωση. Και μετά έδωσαν λαβή, όπω μα είπε και πριν από λίγο ο κύριος Τζάρμαν, και έδωσαν λαβή για μια ευρεία κλίμακα καταστολή τη κοινωνία των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Ε, στόχο έχουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα εκφοβισμού και τρόμου σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Ρωσίας. Δεν μπορούμε να μιλούμε για κράτο δικαίου όταν κυριαρχεί η αυθαιρεσία και ο φόβο, ακόμη και στο δικαστικό μηχανισμό. Δυστυχώ η κρίση έδειξε ότι η απελευθέρωση που είδαμε πρόσφατα δεν ήταν παρά μια απλή ανοχή, ένα διάλειμμα, μια πρόσωψη, μια απλή παρένθεση, χωρί να αμφισβητείται η λογική ενό αυταρχικού ιδιαίτερα κεντρικού συστήματο, χωρί να εξασφαλίζεται η ειρηνική άσκηση ή απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους πολίτες και η απονομή χάρητος από τον πρόεδρο μετά από βεβαιασμένες ομολογίες ή ψευδομαρτυρίες ή συνοπτικές δίκες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την απέτηση δικαιοσύνης και αλήθειας. Όλα τα υπόλοιπα θα ήταν απλώς κάποιοι διπλωματικοί χειρισμοί. Η παρούσα κρίση δεν αφορά μόνο τη Λευκορωσία, ούτε καν τις γειτονικέ χώρες, αλλά θέτει ένα αφιβόλο το σύνολο των αρχών και των δεσμεύσεων ε, και των δημοκρατικών αρχών που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρώπης. Μία μόνη βιώσιμη λύση θα ήταν μία ρηξικέλευθη μετα... μεταρρύθμιση προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κράτος δικαίου με βάση τη διάκριση των εξουσιών, το σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών, τη ελευθερία του συνέρχεσαι μεταξύ άλλων και τη ελευθερία έκφραση, μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαιοσύνη, ε, ένδικων μέσων και διεθνών εγγύσεων. Η έκθεση περιλαμβάνει και μια σειρά συγκεκριμένων και ρεαλιστικών συστάσεων που μπορεί να επιτρέψουν στη Λευκορωσία να ξεφύγει από αυτό το διέξοδο με στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα στα πλαίσια της ΟΑΣΕ αλλά και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από την άποψη αυτή, ο μηχανισμό τη Μόσχας δεν είναι αυτοσκοπό. δεν είναι παρά μόνο ένα στάδιο, ένα σημείο αφετηρία, μια έκκληση ανάληψη ευθυνών και έκφραση πολιτική βούληση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστατεί σε αυτή την συλλογική κινητοποίηση. Τα γραφεία, το, το Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο ΝΤΙΡ, θα πρέπει να προβεί σε μια αξιολόγηση των διαφόρων αυτών δικαίων όταν, όταν ολοκληρωθούν αυτά τα ζωφερά σενάρια και θα πρέπει να... Ε, ε, η Λευκορωσία έχει καταγγείλει την άχρηστη κατά τη γνώμη της προσφυγής στο μηχανισμό της Μόσχας αλλά ε, ο Οντίρ έκλεισε δυστυχώς, έκλεισε μάλλον το γραφείο του ΜΙΣΚ στα τέλη του 2010 στο ΜΙΣΚ. Όπως ξέρετε και το ψήφισμα της 16ης Ιουνίου του 2011 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με μία ψήφους υπέρ, 5 κατά και 19 αποχές αναθέτει στον ύπατο αρμοστή των Ηνωμένων Αθηνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα να υποβάλει μια πρώτη έκθεση για την εξέλιξη της κατάστασης στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει το Σεπτέμβριο και ζητά από τους θεματικούς εισηγητές να μεριμνήσουν για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόπου. Η Λευκορωσία δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να ε, εφαρμόζει καταστολή και καταπίεση ως μόνη απάντηση του καθεστώτος σε μια όλο και πιο οξία και δεινή κοινωνική κρίση. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος ε, Μπιαλιάτσκι. Ευχαριστώ. Όλοι έχουμε αναρωτηθεί γιατί η κυβέρνηση και οι αρχές ε, ε, έδειξαν τόσο στιγμή καταστολή ε, στη διαδήλωση αυτή. Απάντηση δεν έχουμε ακόμα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό προκλήθηκε από το απροσδόκητο του γεγονότος. Ε, δεκάδες χιλιάδες πολιτών ε, κατέβηκαν στη διαδήλωση αυτή και η κυβέρνηση και οι αρχές ήθελαν να καταστήλει την έκφραση αυτή της δυσφορίας και της έλλειψης ικανοποίησης του πληθυσμού. Ήταν ένα τμήμα της μαζικής καταστολής που ακόμα συνεχίζεται και σήμερα. Αυτό το λένε ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί ακτιβιστές. Είναι μια καταστολή και μια καταπίεση χωρίς τέλος. Δεν υπάρχει δυνατότητα βέβαια αντιμετώπισης ε, της ε, αντιπολίτευσης εν μία νυχτή. Δεν μπορούν να την ε, καταστήλουν σε μία νύχτα. Γι' αυτό έχουν ένα ολόκληρο σχέδιο. Η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ ενεργή. 50% ο πληθυσμός, τους ο πληθωρισμός, συγγνώμη, τους τελευταίους τρεις μήνες και υποχρεώνει τις αρχές της χώρας να ε, έχουν απέναντί τους ε, όχι απλώς κάποιους μεμονωμένους πολιτικούς ακτιβιστές, αλλά ολόκληρο το, μάζα εντό εισαγωγικών του πληθυσμού των Λευκορώσων. Η πλειονότητα των Λευκορώσων σήμερα ζει στη φτώχεια και η δημοτικότητα του Λουκασέγκο πέφτει μήνα με το μήνα. Η οικονομική κρίση συνδέεται και με τη μείωση της οικονομικής υποστήριξης από τη Ρωσία. Τα τελευταία τρία χρόνια διαπιστώνεται κάποια μείωση της οικονομικής ε, υποστήριξης από τη Ρωσία. Έπεσε στο μισό και ο σημερινός πρωθυπουργός της Ρωσίας, Πούτιν, δίνει 5 δισεκατομμύρια δολάρια ε, στη Λευκορωσία το χρόνο. Δεν αρκεί αυτό όμως στο Λουκασέγκο και ε, στις αρχές της χώρας. Εργάζονται ε, στην κατεύθυνση μια Τελωνιακή ένωσης ε, Ρωσίας, Λευκορωσίας, Καζακστάν για να επικρατούν και στις τρεις χώρες οι ίδιε τιμέ ε, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ταυτόχρονα όμως θέλουν και την ανεξαρτησία τους να τη διατηρούν με δικές τους οικονομικές πολιτικές και οικονομικά μέτρα. Ως αποτέλεσμα λοιπόν της οικονομικής κρίσης έχουν ε, γίνει μαζικές ε, οικονομικές δραστηριότητες. Την δυσφορία τους και τη διαμαρτυρία τους εκφράζουν οι νέοι, κυρίως μέσω του διαδικτύου. Αλλά δεν έχουν αποδέκτες. Τελικά τι γίνεται με αυτές τις διαμαρτυρίες. Ο κόσμος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βγαίνει στους δρόμους και να ε, χτυπάει ρυθμικά τα χέρια του. Παντού, σε όλες τις πόλεις, πολλές διαδηλώσεις και πολλές συλλήψεις. Πάνω από 2.000 πολίτες έχουν συλληφθεί και πάνω από 1.000 καταδικάστηκαν για χολιγανισμό. Απλούστατο. Έχουμε διαπιστώσει και περιπτώσεις που ε, προπυλακίστηκαν οι ε, διαδηλωτές και ε, που συνελήφθησαν από ανθρώπους με πολιτικά. Πολλές φορές τα δικαστηρία δεν κλητεύουν μάρτυρες και δικάζουν συνοπτικά βάσει εγγράφων που τους προσκομίζει η αστυνομία και η κυβέρνηση της χώρας δεν έχει καμία προθυμία να συζητήσει με την αντιπολίτευση. Είδαμε πώς έγιναν οι δίκες κατά των πολιτικών ακτιβιστών. Μέχρι σήμερα πάνω από 40 πολίτες έχουν ε, καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης για δραστηριότητες στις 19 ε, Δεκεμβρίου του 2010. Μερικοί από αυτούς είναι πολύ βαριά ασθενείς. Κανένα κανόνα δεν σέβεται το κράτος ε, σε ό,τι αφορά τη κράτηση πολιτικών κρατουμένων. Και τώρα απευθύνουμε μία έκκληση στους ευρωβουλευτές να μην σταματήσετε να ασκείτε πίεση, να μην χαλαρώσετε την πίεση προς τις αρχές της χώρας. Ο Αντρέι Πατσόποτοφ, ένας δημοσιογράφος, όλης καταδικάστηκε Στη συνέχεια αφέθηκε ε, ελεύθερος. Έκλεισε μια κρατική εφημερίδα, όπως γνωρίζετε, μια, μια κυκλοφορία κυκλοφορίας εφημερίδα. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εξ ονόματος των ακτιβιστών, των αγωνιστών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων για την προσοχή που δίνει στην κατάσταση στη Λευκορωσία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ελπίζουμε προσοχή αυτή να συνεχιστεί και το φθινόπωρο, διότι πιστεύω ότι η κατάσταση θα οξυνθεί. Γι' αυτό αφορά και την πολιτική και την οικονομική κρίση. Θα παρατηρηθεί κλιμάκωση. Επίσης, οι πολίτες, ο μέσος πολίτης ε, Τη Λευκορωσία γνωρίζει ότι είστε στο πλευρό του και θέλουμε να σας ζητήσουμε να μειώσετε και το κόστος για τη θεώρηση διαβατηρίων για τους Λευκορώσους και καταλαβαίνουν οι Λευκορώσοι οι πολίτες τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για πέντε λεπτά ο κύριο Προτάσεβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πολωνικά αν μου επιτρέπετε. Μιμούμενος των ε, αντιπρόεδρο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Γκζίπ. Επαναλαμβάνω, θα μιλήσω πολωνικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ε, προλαλήσαντες, ε, τους εμπειρογνώμονες του πάνελ μας, που είτε με πρωτοβουλίες μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε κράτη-μέλη της ΟΑΣΕ, είτε όπως ο κύριος Δεκό αναλαμβάνοντας εισήγηση, εκπόνηση έκθεσης με εντολή του ΟΣΕ έχουν πολύ σημαντικό έργο και πολύ σημαντικό είναι και για μας. Όπως θα θυμάστε, εμείς από την αρχή, από το Δεκέμβριο δηλαδή του 2010, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, ε, εκ μέρους του Προέδρου του κ. Μπούζεκ αλλά και η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία εκφράσαμε ε, μία, ένα περίφραστο και στεναρό μήνυμα καταδικάζοντας τα επεισόδια της, ε, του Δεκεμβρίου του 2010 αλλά και τα συμβάντα που ακολούθησαν μετά το Δεκέμβριο. Η αντίδρασή μας όμως ε, πώς ερμηνεύθηκε από τις λευκορωσικές αρχές. Συνεχίστηκαν οι κατηγορίες εις βάρος μας ότι είμαστε ε, υποκειμενική, ότι μεροληπτούμε, ότι είμαστε στο πλευρό της ε, λευκορωσικής αντιπολίτευσης και επίσης είμαστε ριζοσπαστικοί ε, σε ό,τι αφορά την ερμηνεία της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εσωτερικής κατάστασης που επικρατεί και μας κατηγόρησαν και για πολιτικά φελής και αντιπαραγωγικούς. Όλες αυτές ήταν οι κατηγορίες που μας εξακόντισαν οι λευκορωσικές αρχές. Ποια ήταν η δική μας απάντηση. Εμείς συζητήσαμε με τους διπλωματικούς μας εταίρους που εκπροσωπούσαν επίσημα το ΜΙΣΚ ότι δεν ήμασταν εμείς, ε, δεν ήταν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αποστολή μας που έκρινε ως ε, έκρινε τις λευκορωσικές εκλογές ως ε, μη δημοκρατικές και ελεύθερες αλλά η αποστολή της ΟΑΣΕ στην οποία συμμετέχει ε, και η Λευκορωσία εξέδωσαν αυτή την ετοιμικόρια ότι οι εκλογέ στη Λευκορωσία δεν ήταν ελεύθερε και δημοκρατικέ ή ανώθευτε. Εμεί διαπιστώνουμε καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίση παραβίαση των στοιχειωδών προδιαγραφών των δημοκρατικών θεσμών, των ελευθεριών των πολιτών, των ελευθεριών της, της, των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Διαπιστώνουμε καταστρατήγηση αυτών των στοιχειωδών και θεμελιωδών ελευθεριών. Και οι προσκεκλημένοι μας νομίζω ότι έκαναν μια αντικειμενική αξιολόγηση της κατάστασης και μάλιστα εκ μέρου μια οργάνωση τη ΟΑΣΕ, στην οποία συμμετέχει και η ίδια και η Λευκορωσία. Αυτό είπαμε στου συνομιλητέ μα από τη Λευκορωσία. Γιατί δεν υπογράφετε τα τρία νομικά έγγραφα που έχετε προσυπογράψει. Γιατί αν η ΟΣΕ μιλάει για ανάγκη τήρηση ορισμένων προδιαγραφών, γιατί δεν τις τηρείτε αυτές τις προδιαγραφές. Αυτό περιμένουμε από εσά. Ακούσαμε και ένα άλλο επιχείρημα, ότι η λευκορωσική κοινωνία δεν είναι έτοιμη για τη δημοκρατία. Ότι μετά από κάθε απολυταρχικό καθεστώς και ιδιαίτερα ε, χώρες που έχουν από την άξη το Σοβιετικό ζυγό, έχουν πολύ μακρύ δρόμο προς την ελευθερία και τη δημοκρατία. Είναι πολύ πιο χρονοβόρα για τις κοινωνίες αυτές η διαδικασία ότι θα πρέπει να βρει το δρόμο της η Λευκορωσία μέσω των διαφόρων διεθνών προδιαγραφών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρητικά τουλάχιστον και σε κάποιο βαθμό θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με το επιχείρημα αυτό ότι ορισμένες χώρες, ορισμένες κοινωνίες έχουν πιο μακρύ δρόμο προς τη δημοκρατία από ό,τι άλλες. Και ίσως ο, ο ρυθμός της Λευκορωσίας να μην είναι τόσο γρήγορος όσο της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Λιθουανίας, της ε, Ουγγαρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμη και με αργό ρυθμό θα έπρεπε η κατάσταση να αλλάξει, όπως έγινε στην Ουκρανία. Διαπιστώνουμε όμως ότι στη Λευκορωσία όχι μόνο δεν υπάρχουν ελευθερίες, όχι μόνο δεν υπάρχει προσέγγιση των δημοκρατικών αρχών και αξιών, αλλά αντίθετα υπάρχει παλινοδία, επιδείνωση της κατάστασης. Υπάρχουν και μερικές παρανοϊκές και ίσως ε, είναι αυστηρός ο χαρακτηρισμός, αλλά γίνονται παρανοϊκές ε, ενέργειες και μερικές φορές γίνονται συλλήψεις ανθρώπων που απλώς περπατάνε ελεύθερος στους δρόμους, ούτε καν ε, κραυγάζουν, ούτε καν σηκώνουν ε, συνθήματα ή ταμπέλες, απλώς προχωράνε στους δρόμους, μπορεί να χτυπάνε τα χέρια τους, αλλά ακόμη και γι' αυτό ε, συλλαμβάνονται και περνάνε στο κρατητήριο μέρες ολόκληρες. Αυτό όχι μόνο είναι αντιδημοκρατικό, αλλά είναι πραγματικά μία αλλοπρόσαλη παρανοϊκή συμπεριφορά εκ μέρους των λευκορωσικών αρχών. Νομίζω ότι αυτό αφορά ε, περίπου 170 άτομα που υπέστησαν αυτή τη στιγμή καταπίεση και καταστολή. Είναι περιπτώσεις ε, αστυνομικής βίας και σύλληψη αθώων πολιτών που δεν έκαναν τίποτα, απλώ περπατούσαν ελεύθερου στου δρόμου. Και μάλιστα μία γυναίκα που δεν συμμετείχε καν στη διαδήλωση, απλώ τυχαία περνούσε από εκείνο το, το σημείο και ήταν και έγκυο. Υπέστη την ε, στιγμή καταπίεση εκ μέρου των αστυνομικών αρχών και νομίζω ότι απέβαλε κιόλα η γυναίκα αυτή. Έχασε το παιδί της. Επίσης μιλήσαμε για την ε, καταπίεση των, ε, μαζικών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρακτηριστική περίπτωση του Αντζέι Ποτσεμπούτα, ε, Πολωνού δημοσιογράφου, που βρέθηκε με νόμιμα διεπιστευτήρια, νόμιμα προς, έχει προσληφθεί στη Λευκορωσία, από πολωνική εφημερίδα και μάλιστα συνελήθη καταδικάστηκε σε τρίμηνη φυλάκιση και κάναμε διάφορα διαβήματα και μάλιστα για τρεις ε, μήνες έμεινε σε προφυλάκηση χωρίς καμία απαγγελία κατηγορίας και παρά τα διαβήματα που κάνουμε ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε επαφή μαζί του. Ε, τελικά εγκρίθηκαν κάποιες ε, κυρώσεις οικονομικές προς το παρόν Κάτι είναι και αυτό, πολύ μικρό βήμα. Θα ήθελα να αναφέρω ε, τα λόγια ενός διπλωμάτη που τελικά που είπε ότι τελικά οι κυρώσεις έφεραν κάποια αποτελέσματα γιατί τουλάχιστον ε, αποφυλακίστηκε ο Αντζέι Ποτσεμπούτα καταδικάστηκε αλλά με αναστολή και νομίζω ότι απέναντι στο λευκορωσικό καθεστώς οι κυρώσεις είναι το μόνο ε, εργαλείο που έχουν στο, στα χέρια τους, ε, που έχει στα χέρια της Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Παλέτσκι, στον εισηγητή της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή η πολιτική και οικονομική κρίση η οποία διανύει ε, η Λευκορωσία εδώ και έξι μήνες και πλέον αποτελεί ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει και να προωθήσει το δικό της όραμα. Μια Λευκορωσία ανεξάρτητη, δημοκρατική, που είναι γείτονά μας και που θα εφαρμόζει την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Από την άλλη βέβαια είναι σαφές αυτό που τόνισε ο εμπειρογνώμων μας, ότι οι Βρυξέλλες δεν μπορούν να επιστρέψουν στον περιορισμένο διάλογο με το Μίνσκ που ε, ίσχυε πριν τη 19η Δεκεμβρίου εκτός εάν αφαιθούν ελεύθεροι και οι 40 πολιτικοί κρατούμενοι και έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους. Ακούμε κάποιες ειδήσει ε, σχετικά, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούμε πολύ ε, κοντά την κατάσταση για να δούμε τι όρους και προϋποθέσεις μπορούμε να θέσουμε αν μπορούν κάποιοι να αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά τονίζω ότι θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, που είναι πάνω από 40. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ε, συνεργαστεί περισσότερο με την Ουκρανία και τη Ρωσία για το θέμα αυτό. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ε, συναντηθήκαμε με τον Κωνσταντίν Γκρισέγκο, ε, Ουκρανό Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και το ρώτησα τι κάνει το Κίεβο για όλα αυτά. Και απάντησε ότι η κυβέρνηση εργάζεται ε, σκληρά και συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Λευκορωσίας και πιέζει το Μίνσκ να φέρει σε ελεύθερους πολιτικούς κρατουμένους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το μήνυμα αυτό. Βεβαίως, έχει ιδιαίτερη σημασία πάντα να καταλάβει η Μόσχα ότι ο εξυγχρονισμός ε, της εταιρική της σχέσης με την ε- Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την πολιτική και οικονομική εξέλιξη και τον εξυγχρονισμό γειτονικών μας χωρών και των δύο όπως είναι η Λευκορωσία. Επίση τονίζεται η ανάγκη να βελτιωθεί ε, το σύστημα και το καθεστώ θεώρηση διαβατηρίων για τους λευκορώσους πολίτες. Επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο έχουμε τονίσει ότι έχουμε ορθώσει ένα νέο τείχο του Βερολίνου, οικονομικό, για το μέσο πολίτη της Λευκορωσίας που θα πρέπει να καταβάλει το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο του μισθού του για να πάρει βίζα για ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περασμένη εβδομάδα μια γερμανική επιτροπή ε, για τις σχέσεις με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, ε, τις οικονομικές, εξέδωσε μια μελέτη 200 ε, εταιριών ακριβώς για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και γύρω στο 25% ε, των εταιριών χάνουν τα συμβόλαια και τις ε, εμπορικές τους συναλλαγές γιατί δεν παίρνουν θεώρηση διαβατηρίου να κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Και ελπίζω αυτά να μην είναι θέματα του αποτέρου αλλά του προσεχούς μέλλοντος. Και ένα τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως θα πρέπει να εντείνει τη συνεργασία της με την αντιπολίτευση στη Λευκορωσία, όπως και πράττουμε άλλωστε. Και από την άλλη θα ήταν χρήσιμο να αναζητήσουμε επαφές με ε, μετριοπαθείς πολιτικούς και στο Μίνσκ και αλλού, στις πόλεις, στα χωριά και με στελέχη του σημερινού καθεστώτος. Διότι και εκείνοι θέλουν ορισμένοι να δουν και αλλαγή καθεστώτος και μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Θα παρακαλέσω τον κύριο Βιγγένιν που είναι συμπρόεδρος ε, της ε, Euronest, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ε, Θα ήθελα να σας πω ότι η σημερινή ε, συζήτηση ε, γίνεται με μια αρνητική αφορμή τις προεδρικές εκλογές. Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, που όχι το αποτέλεσμα, το πω ο τερματισμός των προεδρικών εκλογών ήταν απογοήτευση. Πριν τις εκλογές θεωρούσαμε ότι άρχισε σιγά σιγά η κατάσταση να βελτιώνεται. Η ημέρα όμως της εκλογικής αναμέτρησης εξελίχθηκε πάρα πολύ διαφορετικά. Ε, στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής συνέλευσης Euronest, που συνεδρίασε αρχές ε, Μαΐου και συστήθηκε σε σώμα, απουσία της Λευκορωσίας, πρέπει να πούμε ότι ήταν μια παρένθεση εδώ. Ε, θέλαμε να συμμετέχει η Λευκορωσία, ήταν τελείω αδύνατο μετά τι προεδρικέ εκλογέ. Κλείνει η παρένθεση. Εκεί λοιπόν στη Euronet συστήθηκε μια ομάδα ε, για τη Λευκορωσία που απαρτίζεται από εκπροσώπου ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από τις υπόλοιπες πέντε βουλές των κρατών της Ανατολικής Γειτονίας. Αυτή η ομάδα εργασίας έχει δύο προέδρους, ένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα από τη Μολδαβική Βουλή. Αυτή η ομάδα εργασίας φιλοδοξεί να καθιερώσει μια συνεργασία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ε, γειτονές μας ε, ξανατολών, την Ουκρανία για παράδειγμα. Και με κάποιο τρόπο να μπορεί να συμμετέχει, ή να πρέπει να συμμετέχει και η Ρωσία πιστεύουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά τη Λεύκο πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία εκεί. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι του προσκεκλημένου μας τους προσκεκλημένους μας που γνωρίζουν την κατάσταση και παρακολουθούν τις εξελίξεις ε, από πολύ κοντά στη Λευκορωσία. Έχω την εξής λοιπόν ερώτηση. Υπάρχουν πιθανότητες στη Λευκορωσία να επικρατήσει ελευθερία κάποια στιγμή και ποιες είναι αυτές, πόσες πιθανότητες. Και όταν μιλώ για ελευθερία εννοώ ελεύθερες εκλογές με βάση τα διεθνή πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με τη σειρά της πιστεύω έχει περιορισμένες δυνατότητες να παρέμβει. Νομίζω ότι έχουμε ήδη κάνει ό,τι περνούσε από τα χέρια μας. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει τις θύρες για τους πολίτες της Λευκορωσίας και προσπαθούμε να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην συνεργασία με το κράτος ε, και με τη συνεργασία που έχουμε με τους Λευκορώσους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, όχι το επίσημο κράτος. Γι' αυτό λοιπόν αν διευκολύνουμε και το καθεστώς θεώρηση διαβατηρίων θα κάνουμε ακόμα ένα βήμα προς την κατεύθυνση των λευκορώσων πολιτών και όχι του καθεστώτος. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την αντιπολίτευση ακόμα περισσότερο υπό την πολιτική αλλά και την ηθική έννοια ενώ την υποστήριξη. για να την ενισχύσουμε, για να τη σταθεροποιήσουμε. Η αντιπολίτευση έρχεται συχνά εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά μετά είδαμε τι μεταχείριση επιφυλάσσει το κράτος ε, στους αντιπολιτευομένους. Το τελευταίο διάστημα είχαμε επεισόδια και συμβάντα που ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι η Λευκορωσία είναι ή μη αστυνομικό καθεστώς. Αυτό θα προκαλέσει επιπλέον δυσκολίες και προβλήματα, αλλά η πίεση δεν θα πρέπει να χαλαρώσει και εσωτερική και εξωτερική και σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική κρίση και νομίζω αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω, τι γνωρίζουμε για τα επεισόδια, τα γεγονότα της 19ης Δεκεμβρίου το 2010 και τι είδαμε. Ο Λουκασένκο και η Κάγκεμπέ του ήταν έτοιμοι να επιτεθούν στους ε, αντιφρονούντες ε, γιατί μισούν την πολιτική ε, αντιπολίτευση. Και βρήκαν τώρα μια αφορμή μερικούς που ε, έφτασαν κοντά σε ένα κτίριο και είχαν φυσική επαφή με παράθυρα και πόρτες. Οι πολίτες έλεγαν ε, «σταματήστε, μην κάνετε τέτοια». Και για να το συγκρίνουμε με άλλες καταστάσεις, ε, όταν οι διαδηλωτές ε, πλησίαζαν απειλητικά το προεδρικό μέγαρο, ο κύριος Μιλικίεβιτς τους έλεγε σταματήστε. Παρόλα αυτά καταδικάστηκε αργότερα ε, μεταξύ άλλων προσωπικότητων αυτής της ενωμένη αντιπολίτευσης. Και τον λένε και προδότη μάλιστα. Διδάγματα έχουν εξαχθεί από όλα αυτά που συνέβησαν ή όχι. Και τώρα υπάρχει καμιά ευκαιρία να συσταθεί και να διατηρηθεί μια ενωμένη δημοκρατική αντιπολίτευση με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και τακτική. Υπάρχει έδαφος. Για κάποιες αιτιάσεις ε, της κυβέρνησης ότι η αντιπολίτευση ε, υποκινείται και από τη Δύση και από τη Μόσχα. Ευχαριστώ. Äh, Η ερώτησή μου έρχεται ακριβώς να ε, συμπληρώσει αυτά που είπε ο κύριος Λαντσμπέργης. Αν ήταν προβοκάτορες, αυτοί οι προβοκάτορες έχουν αναγνωριστεί, γιατί είναι και στη τηλεόραση εικόνες, τους βλέπουμε με μονομένους ε, πολίτες που ε, με βία να επιτίθενται σε κάποια κτίρια. Μέχρι τώρα έχω μάθει ότι αυτοί που έχουν συλληφθεί ήταν διαδηλωτέ που δεν είχαν καμία σχέση. Λοιπόν, αν γίνει κανονική έρευνα, αυτού μπορούν να του βρουν. Και η δεύτερη ερώτηση ε, είναι προ τον ε, Αλεξάνδρου Μπιαλέτσκι Ένα τέτοιο πολιτικό μοντέλο όπως η στρογγυλή τράπεζα που είναι στην Πολωνία ή στην Ανατολική Γερμανία ε, θα ήταν ευκαιρία για τη Λευκορωσία. Δηλαδή διαπραγματεύσεις από τη σημερινή ολοκληρωτική κυβέρνηση με εκπροσώπους ε, της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον τους επόμενους μήνες. Κάποια πολιτική συνένεση δεν μπορείτε να βρείτε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ε, πολύ ενθαρρυντικά τα στοιχεία ως προς την ε, ε, κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αρχή της ερεσιμότητας που θα πρέπει να ισχύσει. Δηλαδή, μόνο εάν απελευθερωθούν οι φυλακιστέντες, τότε θα αρχίσουμε ένα νέο πολιτικό διάλογο η κατάσταση ήταν λίγο διαφορετική ένα χρόνο πριν. Και τότε θέλαμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία με το Λουκασέγκο. Αλλά δεν μπορεί κανείς να ε, δέχεται και να εμπιστεύεται τους δικτάτορες. Θα ήθελα να πω στους προσκεκλημένους μας να τους ρωτήσω πώς κρίνεται τα τελευταία ε, γεγονότα και πώς κρίνεται την κοινωνία των πολιτών. Η νέα γενιά χρησιμοποιεί το Facebook, τους υπολογιστές και ούτω καθεξής. Μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους οργανώσεις με αυτόν τον τρόπο. Πώς μπορεί να αποκατασταθεί και να υπάρξει μια ενωμένη αντιπολίτευση. Αυτός είναι ένας ε, απαράβατος όρος και ο Επίτροπος Φούλερ ήρθε σε επαφή με πολλά μέλη της αντιπολίτευσης και τους ενθάρρυνε να ενωθούν, τους προέτρεψε να ενωθούν. Πιστεύω ότι μπορεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει ε, αυτούς τους, ε, τους φυλακισμένους και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κανείς να αναλάβει μια συγκεκριμένη ευθύνη και δράση εναντί των ε, φυλακιστέντων. Η κυρία Αντρικένε, θα μιλήσω στα λιθουανικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να αρχίσω με αυτά που μόλις είπε ο κύριος Πρωτασέβιτς. Πράγματι, είναι γεγονός ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία επιδεινώνεται ένα και περισσότερο. Και αυτό δείχνει και την αδυναμία του καθεστώτος όταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων που συγκεντρώνονται και επιχειροκροτούν στους δρόμους συλλαμβάνονται. Αυτό δείχνει την, την κατάσταση απελπισία στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση και νομίζω ότι το φθινόπωρο θα ε, υπάρξουν εξελίξεις στη Λευκορωσία. Θα ήθελα να υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις προς τον κύριο Μπελέτσκι και στους άλλους παρεμβαίνοντες. Πώς βλέπετε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει μία φωνή, να εκφράζεται με μία φωνή, διότι υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που έχουν μία καθαρά πραγματιστική ε, θέση σε σχέση με τη Λευκορωσία. Ναι, πράγματι, είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι ερωτήσεις και επειδή πρέπει να λήξει ο γύρος, να λήξει η συζήτηση σε ένα τέταρτο, νομίζω ότι θα μπορούσατε να έχετε πέντε λεπτά ο καθένας για να απαντήσετε. Θα πρέπει να αντιστρέψουμε την αρχή και θα αρχίσουμε με τον κύριο Γκαλεάτσκι, μετά ο κύριο Ντεκόν και ο κύριο Γιάνναν. Έχετε το λόγο λοιπόν. Εάν πρόκειται να μιλήσουμε για την έκβαση των ε, εκλογών του ε, χρόνου το φθινόπωρο, γιατί θα διενεργηθούν εκλογές, εάν μπορούν να είναι πραγματικά ελεύθερες εκλογές, αυτό θα ήταν πραγματικά κάτι το απόλυτα επιθυμητό. Όμως, εάν οι αρχές δεν τηρήσουν τους όρους που θέσατε εσείς για τη διενέργεια των εκλογών, τότε θα μπορούσαμε να μην έχουμε αίσιο πέρας. Μιλάμε για το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας, το δικαίωμα του συνέρχεστε, το δικαίωμα της σύστασης πολιτικών ομάδων και κομμάτων. Εάν δεν γίνουν όλα αυτά δεν θα έχουμε ελεύθερες εκλογές. Η κατάσταση είναι υποεξέλιξη και θα μπορούσαν να διαγραφούν διάφορα σενάρια. Το φθινόπορο θα προωθήσουμε μια πολιτική ε, εμβέλειας εκστρατεία. Υπάρχει ένα σενάριο, ένα καθαρά ενωτικό σενάριο το οποίο προωθείται. Τώρα για το θέμα κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μία ενωμένη δημοκρατική αντιπολίτευση. Αυτό φαίνεται δύσκολο επί του παρόντος. Δεν υπάρχει ενωμένη αντιπολίτευση. Υπάρχουν ζητήματα επί των οποίων είναι ενωμένη η αντιπολίτευση ως προς την απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων, για παράδειγμα, όμως δεν προβλέπονται κοινέ δράσεις. Θα δούμε τι θα συμβεί το φθινόπωρο. Βλέπουμε τι συνέβη σε χώρες όπως η Τινησία. Αυτό δείχνει ότι αν υπάρχει πραγματική διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης, εάν υπάρχουν μαζικά κίνηματα, τότε μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Δεν έχει σημασία η διάρθρωση της ε, δύναμης της αντιπολίτευσης. Πριν από τρεις ε, μήνες είχα μεταβεί στην Τινησία και είδα ότι πραγματικά οι μεγάλες μάζες έφεραν την αλλαγή. Δεν υπήρχε μία συγκροτημένη ε, αντιπολίτευση. Ως προς την αντιπολίτευση, κατά πόσο έχει ε, υπόκειται στην επιρροή της Μόσχας, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ε, η κυβέρνηση έχει ασκήσει και μεγάλη πίεση στην αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση θεωρεί ότι έχει παγιδευτεί από τις μυστικές υπηρεσίες οι οποίες, οι οποίες την ε, πρόδωσαν. Μιλήσαμε και ε, για στοιχεία προβοκάτσιας, τα οποία δεν έχουν όμως διαπιστωθεί παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τι τους, ε, ε, τις δίκες οι οποίες ε, προχωρούν αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτούς που επιτέθηκαν κατά του κρατικού κτηρίου. Όμως αυτοί που φυλακίστηκαν και προσήχθησαν ήταν απλοί πολίτες οι οποίοι δεν είχαν κάνει τίποτα, ούτε έσπασαν τζάμια, ούτε επιτέθηκαν, ούτε τίποτα. Γύρω, στα 30, γύρω στους 30 ήταν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν, ενώ οι συγκεντρωθέντες, οι διαμαρτυρίες ήταν γύρω στους 20 με 30 χιλιάδες. Δεν υπάρχουν λοιπόν αποδεικτικά στοιχεία και οι αρχές της Λευκορωσίας δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένες να διαπραγματευτούν με την αντιπολίτευση. Δεν νομίζω ότι η οικονομική κρίση είναι τόσο, ε, τόσο στεναρή έτσι ώστε δεν έχει πλήξει τόσο πολύ το λαό έτσι ώστε να πρέπει να ε, έρθει σε επαφή η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση, δηλαδή να υποχρεωθεί να προωθήσει ένα διάλογο με την αντιπολίτευση. Νομίζω ότι τους τελευταίους έξι μήνες είχαμε μεγάλες εξελίξεις ως προς την ε, δράση της κοινωνίας των πολιτών. Οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι, οι πολίτες είναι ιδιαίτερα δραστήριοι. Προωθείται αυτή η, ε, η δράση που καλύπτει ένα και μεγαλύτερα στρώματα πολιτών και το κοινό συμμετέχει σε αυτό το κίνημα. Υπάρχουν δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και το κοινό γενικότερα, το οποίο μπόρεσε να αντισταθεί παρά τις πολιτικές δίκες. Ως προσθέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς ακούμε μία φωνή, τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία και εισακούεται και πιστεύω ότι τη στιγμή που υπάρχουν στοχοθετημένες κυρώσεις αυτό αποτελεί ένα πολύ ισχυρό μήνυμα που αποστέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κυβέρνηση της Λευκορωσίας. Αυτό το μήνυμα ελήφθη από την κυβέρνηση και πιστεύω ότι οι πολιτικές πιέσεις και οποιοδήποτε πολιτικός μηχανισμός που ασκεί πίεση προς την κυβέρνηση του Λουκασένκο θα μπορούσε να αποδώσει. Δεν έχει αποδώσει ακόμα και νομίζω ότι μόνο με οικονομική πίεση και κυρώσεις θα μπορέσει να ανταποκριθεί η κυβέρνηση. Ευχαριστώ καθηγητής Δεκό. Πιστεύω καταρχήν ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η αποφυλάξη των πολιτικών κρατουμένων. Όχι μόνο η απελευθέρωση τους όμως, αλλά και η αποκατάστασή τους και η ε, πλήρης ε, άσκηση των δικαιωμάτων τους. Τέθηκε μία ερώτηση για το κλίμα ελευθερίας. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι των ακτιβιστών και υπερμάχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, οι δημοσιογράφοι, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δεν έχουν καταχωρηθεί ε, υφίστανται συνεχώς αυτό το φόβο της απειλής νέου κύματο καταστολών, παρόλο που υπάρχει μια φαινομενική ανοχή απέναντί του. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το βάρος των μυστικών υπηρεσιών της ΚΑΚΕΜΠΕ, που έχει κρατήσει και την ονομασία της. Επίσης, και τις παρεμβολές ε, στο δικαστικό μηχανισμό και το κλίμα τρόμου και φρίκης που επικρατεί με μαύρες λίστες, τα έγιναν ανακρίσεις των παιδιών αντιφρονούντων στα σχολεία τους. Έχουμε λίστες μαύρες ε, με φοιτητέ συγγενείς αντιρρησιών, αντιφρονούντων που δεν μπορούν να φοιτήσουν Υπάρχουν διάφορα τέτοια μέτρα καταστολής και όταν μιλούμε για δικαιοσύνη και δίκες ε, επικρατεί πραγματικά μια θερεσία ακόμη και στο δικαστικό μηχανισμό, ακόμη και για τους δικαστές, γιατί και οι δικαστές αισθάνονται φόβο και οι δικηγόροι ε, δεν μπορούν να υπερασπίσουν ε, τους πελάτες τους κανονικά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μερικά χαρακτηριστικά κομμουνιστική δικτατορία για να καταλάβουμε το κλίμα. Τώρα, ω προς την ουσία, το σημαντικό είναι να μιλάμε ενιαία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσπαθήσει επίση να κινητοποιήσει και του συμμάχου τη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είναι ε, ευαισθητοποιημένε. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να κινητοποιήσουμε όμω και τη Ρωσία και την Ουκρανία και επίσης να βρούμε στοχευμένες έξυπνες κυρώσει που δεν θα κόβουν τελείως επαφές, δεν θα επιδεινώνουν την ίδια επισφαλή οικονομική κατάσταση των πολιτών με κίνδυνο να έχουμε μια νέα κούβα που θα υποστεί μια οικονομική ασφυξία και θα βρεθεί σε κατάσταση οικονομικού αποκλεισμού και πολιορκίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να πολλαπλασιάσουμε τις επαφές και με εκπροσώπους ε, της κυβέρνησης, γιατί δεν είναι κατά ανάγκη όλοι οι φερέφανα του Προέδρου, παρόλο που υπάρχει ένα σύστημα καταστολής επίσημο και στέρεο, παρόλα αυτά υπάρχει και αρχή της, ε, του ρεαλισμού που μερικές φορές την επιβάλλει η οικονομική κρίση. Θα πρέπει να βρούμε μια ε, ήπια μετάβαση και μια αλλαγή. Γνωρίζοντα ότι το λαό δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε όπως έλεγε ο Μπρέχ, θα πρέπει να βρούμε μια βιώσιμη εναλλακτική λύση που θα περάσει κάπου μια πολιτική συμφωνία. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Ο κύριος Τζάρμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το θέμα των πολιτικών κρατουμένων τονίστηκε και είναι ακριβώς πολύ υψηλή προτεραιότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει. Ε, μιλήσατε για την ανάγκη αποκατάστασης, αλλά θα πρέπει πλήρως να εξεταστούν ε, όλες οι κατηγορίες να μην έχουν ποινικό μητρό οι άνθρωποι ότι έχουν καταδικαστεί για ε, ποινικά δικήματα. Θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι ε, να μπορούν να συνεχίσουν τη δράση τους στην κοινωνία. Θα πρέπει πλήρως να διαλευκανθεί η κατάσταση ε, και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καταδικάστηκαν αρχικά. Το θέμα της δικαιοσύνης και της απάντησης που έδωσε στα γεγονότα της 19ης Δεκεμβρίου είναι σημαντικό εκείνοι που, ενήχαν, που μετήχαν και ενέχοντος τα επεισόδια, τα βία, δεν διώχθηκαν. Φαίνεται υπάρχουν στοιχεία, ε, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι ήταν και θα πρέπει να βεβαιωθούμε για ταυτότητά τους και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Χρειάζεται ευρύτερη έρευνα ως προς τις ευθύνες αυτών των πράξεων. Ποιος έδωσε τις ε, διαταγές επέμβασης, ποιος όρισε το χρονικό ε, σημείο που επενεύει η κρατική μηχανή και από ποιο επίπεδο ξεκίνησαν οι δολές και οι διαταγές, από επίπεδο του Προέδρου ή χαμηλότερο. Επίσης, φαίνεται ότι συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες με πολλούς τρόπους και πολύ εφάνταστος, με ε, πολλούς, από πολλούς πολίτες και οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Συχνά υφίστανται κυρώσεις, αστυνομική ε, επέμβαση, ε, διώξεις, συλλήψεις, αλλά φαίνεται όπως έγινε και στη Νότια Μεσόγειο όταν Άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου στις 19 ε, Δεκεμβρίου συγκεκριμένα. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει πίσω το ποτάμι. Έχει φύγει ο φόβος και η αδράνεια. Συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται και η αντίσταση και η αντίδραση και οι διαμαρτυρίες και οι ε, αντιστάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συμμετέχει. Ακούστηκε κάτι για στρογγυλή τράπεζα. Αλλά νομίζω πιο αποτελεσματικό διάλογο, πιο έντονο με την κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία για να καταλήξουν σε μια συμπεφωνημένη λύση, όχι μεταξύ ολίγων, θα ήταν χρήσιμο. Και έτσι μπορούσε ακριβώ να υποστηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, να την αναγνωρίσει, ότι συνεχίζεται δηλαδή και όπω επίση ακούσαμε, μπορεί να υπάρχουν διστάμενες απόψεις και διάφορες φωνές που να ακούγονται, αλλά χρειάζονται υποστήριξη τους επόμενους μήνες. Ο δρόμος θα είναι μακρύς, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω έχει ε, τη δύναμη να πιέσει και τις αρχές και να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υποστηρίζει τις ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών στην καθημερινή τους και συνεχιζόμενη δράση. Ευχαριστώ πολύ ο Αντζέι Γκζίπ και ο κύριος Πρωτοσέβης για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμότατα τους προσκεκλημένους μας ε, για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. και για την νομική ερμηνεία αυτών των ε, επεισοδίων που έλαβαν χώρα στη Λευκορωσία μετά τις 19 Δεκεμβρίου του 2010 και ο κύριος καθηγητής Ντεκό και ο κύριος Τζάρμαν ε, ως εκπρόσωποι διεθνών οργανώσεων μας έδειξαν και μας παρουσίασαν ε, το υπόβαθρο αυτών των ε, συμβάντων, των γεγονότων, την διεξαγωγή τους, την αντίδραση των αρμόδιων αρχών. Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι παρουσιάσεις γιατί αυτή η φιλιρινική διαδήλωση καταστάλει με στιγνό ε, και βίο τρόπο υπό το πρόσχημα καταστολής ε, μιας ε, προβοκάτσιας που έγινε από κάποιες ταραξίες. Είχαμε επίσης φυλάκιση πολλών μελών της αντιπολίτευσης, αντιφρονούντων και το η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να εξασφαλιστεί η αποφυλάκησή τους και φυσικά η ηθική τους αποκατάσταση. Υπάρχει και μια επιβεβαίωση από την ΟΑΣΕ και όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως μας επισήμανε πολύ σωστά ο κύριος Πρότασεβιτς, ο πρόεδρος αντιπροσωπείας για τη σχέση με τη Λευκορωσία. Δεν ήταν μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ε, αισθάνεται αυτή τη δυσφορία απέναντι στις λευκορωσικές αρχές. Και αισθάνεται αποτροπή για τον κατασταλτικό μηχανισμό που εφαρμόζουν οι λευκορωσικέ αρχές. Είναι σημαντικό που και άλλη διεθνή οργάνωση όπω η ΟΑΣΕ έκανε μελέτη και κατέληξε συμπεράσματα παρόμοια με αυτά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε αντιδράσει από την παγκόσμια κοινότητα και να ασκήσουμε πιέσεις για αποφυλάκηση των αντιφρονούντων για δημιουργία ενός συστήματος που θα στηρίζει την κοινωνία των πολιτών και να κινητοποιήσουμε διάφορους μηχανισμούς και εργαλεία προκειμένου η παγκόσμια κοινότητα να ασκήσει πιέσει στις λευκορωσικές αρχές για να εγκριθούν και να εφαρμοστούν κάποιε μεταρρυθμίσει. Σίγουρα δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος και θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρακολούθηση τη περαιτέρω κατάσταση και των γεγονότων που θα ακολουθήσει στη Λευκορωσία. Ο κύριο στα αγγλικά. Θα ήθελα κι εγώ να σε χαρώ και να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας και όλους τους συναδέλφους βουλευτές που μίλησαν για τη συνεισφορά τους, που αν μου επιτρέπετε, συμφωνώ μαζί τους. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τη διεθνή πίεση επί του καθεστώτος της Λευκορωσίας, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να τους αναγκάσουμε να αφήσουν ελεύθερους τους κρατουμένους και ίσως τελικά να προβούν και σε κάποιες αλλαγές ε, για να είναι η κοινωνία πιο ελεύθερη και πιο δημοκρατικό το σύστημα στη χώρα. Ερχόμενος εδώ στη συνεδρίαση μιλούσα στο τηλέφωνο με τον Αντζέι Πότσοβουτ, τον ε, δημοσιογράφο που ε, μόλις αφέθηκε ελεύθερος πριν από λίγες μέρες ε, με αναστολή είχε συλληφθεί προτριμήνου ε, για περίβριση του Προέδρου της χώρας και μου είπε πες σε όλους εκείνους που συμμετέχουν στην ακρόαση ότι με άφησαν ελεύθερο μόνο και μόνο επειδή υπήρξε διεθνής πίεση και οικονομικές κυρώσεις εισήχθησαν και ε, Ε, υπάρχει ακόμα η απειλή των κυρώσεων ότι θα παραταθούν και θα επιβληθούν. Τέτοια μόνο επιχειρήματα καταλαβαίνουν στο Μίνσκ οι αρχές. Γι' αυτό ε, θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και να σας ζητήσω να είστε αμετακίνητοι στη θέση σας, γιατί έτσι θα βελτιωθεί η ζωή των πολιτών της Λευκορωσίας. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ε, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε τους προσκεκλημένους μας και όλου εσά που συμμετείχατε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Thank you very much.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 Please, Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα σας παρακαλώ να καθίσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε τις συζητήσεις μας. Όπως γνωρίζετε το επόμενο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης της Συρίας για την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία μαζί με την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες μας. Θα θέλαμε να ε, καλωσορίσουμε τον κύριο Μάριο Ντέιβιτ που είναι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας. Όπως ξέρετε, εδώ και τρεις ε, μήνες γίνονται διαδηλώσεις στη Συρία, ειρηνευτικές διαδηλώσεις, οι οποίες καταστέλλονται βία από το καθεστώς, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Και την προηγούμενη εβδομάδα, μέσω ψηφίσματος, ζητήσαμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να καταδικάσει τη βία αυτή καταστολή και τις παράνομες ε, φυλακίσεις και κρατήσεις. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τη βία και επέβαλε ε, σοβαρές κυρώσεις. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε για να αποτιμήσουμε την κατάσταση Ε, μέλη της αντιπολίτευσης στο καθεστώς ε, της Συρίας, τον δόκτορα Χαϊτάμ Αλμαλέχ, ο οποίος μόλις ε, απελευθερώθηκε από τη φυλακή το Μάρτιο μετά από 17 μήνες παράνομης κράτησης. Και θα θέλαμε επίσης να καλωσορίσουμε τον κύριο Μπουράν Γκαλιούν, που είναι ο διευθυντής του Κέντρου Μελετών, ε, για, του Κέντρου Μελετών στο Παρίσι για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα ήθελα να ζητήσω από τον δόκτωρα Μαλέχ να μας παρουσιάσει την κατάσταση καταρχήν και θα ήθελα να περιοριστείτε στα 10 λεπτά έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε συζητήσεις. Έχει, το λόγο πρώτα ο κύριος Χαϊταμαλ Μαλέχ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλες τις ε, κυβερνήσεις οι οποίες με βοήθησαν κατά την περίοδο της κράτησής μου κατά την περίοδο της φυλάκισής μου, διότι χρησιμοποίησαν κάθε μέσο για να με βοηθήσουν, έτσι ώστε η κυβέρνηση, το καθεστώς, να με απελευθερώσει. γνωρίζετε την μεγάλη επανάσταση η οποία φαίνεται να εδρεώνεται πλέον στη Συρία. Άρχισε εδώ και τρεις μήνες. Και ε, δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα στιγνό καθεστώς. Από την αρχή της επαναστατικής αυτής δράσης το καθεστώς άρχισε να πυροβολεί τους άοπλους, τους πολίτες, οι οποίοι δεν φέρουν όπλα βεβαίως. Όλοι οι πολίτες της πόλης, τα χωριά, στις κομοπόλεις ε, προέβαιναν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί το καθεστώς ε, πυροβόλησε κατά αυτών των ανθρώπων και σκότωσε πολλούς. Το καθεστώς αυτό από το 1980, από την ε, περίοδο του, του Ασάντ, δεν άλλαξε τίποτα. Μεταξύ ε, 80 και 90, κατά την δεκαετία δεκαετία του 80 χάσαμε 70.000 ανθρώπους με σφαγές, στις φυλακές απεβίωσαν και ούτω καθεξής. Άρα η ίδια λογική διέπει και αυτό το ε, καθεστώς. Δηλαδή ο, ο γιος του Ασάντ, ο Ασάρ, ε, Μπασάρ, ε, δυστυχώς ε, ακολουθεί την ίδια λογική. Εμείς ως αντιπολίτευση Ζητήσαμε από το καθεστώς να προβεί σε διάλογο, να ξεκινήσει ένα διάλογο, να σταματήσει τις δολοφονίες. Να απομακρυνθούν τα τάγκς και να σταματήσουν οι επιθέσεις από τις μυστικές υπηρεσίες, να μην χρησιμοποιεί τη στιγμή αυτή η δύναμη για να σταματήσει την επανάσταση και να μας ε, επιτρέπει να συγκεντρωθούμε έτσι ώστε να συζητήσουμε και να αποτιμήσουμε την κατάσταση. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Δυστυχώς συνεχίζονται οι φυλακίσεις, οι προσαγωγές, οι δολοφονίες και τώρα κρατούνται στις φυλακές 15.000 πολίτες και για κανένα λόγο. 2.000 είναι οι σκοτωμένοι και 500 είναι αγνοούμενοι. Περίπου 100 παιδιά κάτω των 15 ή των 12 έχουν εξαφανιστεί και δημιουργούνται, μάλλον χρησιμοποιούνται τα βασανιστήρια, τα στιγνά βασανιστήρια, ενώ θα έπρεπε να σταματήσουν στη χώρα. Το καθεστώς αυτό δεν ε, τιμά τις υπογραφές του στις διεθνείς συμβάσεις. Δεν τιμά την υπογραφή του, το λόγο του. Δεν τηρεί το νόμο, το γράμμα του νόμου, οποιοδήποτε νόμου. Κυβερνεί με διατάγματα. Δυστυχώς ο νόμος αποτελεί νεκρό γράμμα. Άρα καταλαβαίνετε πώς μπορούμε να, να επιζήσουμε και να διαβιώσουμε κάτω από αυτό το καθεστώς. Ε, εγώ έστειλα πολλές επιστολές στον Μπασαράσαντ από την αρχή του καθεστώτος του εδώ και δέκα χρόνια και σε πολλούς άλλους υπουργούς, τις μυστικές δυνάμεις, ήρθα σε επαφή με πολλούς αξιωματούχους, όμως δεν συνέβη τίποτα. Βλέπουν λοιπόν οι πολίτες ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διαλόγου. Όπως σας είπα, ε, είχαμε, γνωρίσαμε μεγάλη αιματοχυσία Βεβαίως το καθεστώς δεν το απασχολεί αυτό. Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής και από τη δική μας πλευρά, η αντιπολίτευση δηλαδή, προσπάθησε να οργανώσει ορισμένες συγκεντρώσεις για να συζητήσουμε για το μέλλον της χώρας. Γιατί πιστεύουμε ότι το καθεστώς αυτό έχει αποτύχει, έχει τελειώσει. δεν μπορεί να κυβερνά πλέον. Κατά την άποψή μου αυτό το καθεστώς ε, ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Δεν τηρεί το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημοσιεύει νέους νόμους για να κυβερνά τη χώρα. Θα πρέπει να αποχωρήσει και να μας αφήσει να αλλάξουμε το πρόσωπο αυτής της χώρας. Δηλαδή να περάσουμε από την ε, δικατατορία στη δημοκρατία σε μια χώρα ελευθερίας όπου θα τηρούνται τα δικαιώματα, θα την χάνουν σεβασμού δηλαδή τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεπιθήσεις. Στη Δαμασκό στις 16 του μηνός θα συζητήσουμε για το μέλλον της Συρίας, εμείς ως αντιπολίτευση και προβλέπεται και μία συνάντηση στην Ισταμπούλ την ίδια ημέρα με εξωγενείς παράγοντες και τις τελευταίες ημέρες ε, προβλέπεται και μία ε, συνάντηση ολόκληρης της αντιπολίτευσης για να δούμε ποια θα είναι η μελλοντική μας πορεία. Στη Συρία ο λαός πιστεύει ότι η Ευρώπη είναι πραγματικός εταίρος Έχουμε μία μακραίωνη ιστορία σχέσεων με την Ευρώπη και θεωρώ ότι αν η Ευρώπη βοηθήσει την επανάσταση, βοηθήσει το λαό που κινείται πλέον και εκφράζεται στους δρόμους, θα είναι πολύ θετικό και για τις δύο πλευρές και ιδιαίτερα για τους μετανάστες. Ίσως αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις μεταναστευτικές ροές από τη χώρα μας. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι μπορέσουμε να δώσουμε ένα καλό ε, μέλλον, να υπάρξει ένα θετικό μέλλον και θετικές κινήσεις για το μέλλον μας, τότε αυτό θα είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Οι στρατιωτικές δυνάμεις οι ένοπλες δυνάμεις δρούν. Έχουμε 3.000 τάγκ σε ολόκληρη τη Συρία, στη Μπανιάς και γύρω από τη Μπανιάς. Κινούνται οι ένοπλες δυνάμεις με τα τάγκ. Δεν υπάρχει ε, δεν υπάρχει ένομη τάξη, δεν, υπάρχουν, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν είδη διατροφής, αποχωρούν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Δεν υπάρχει υδροδότηση, δεν υπάρχουν τρόφιμα και δυστυχώς απομακρύνονται όλοι από τα σπίτια τους. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη δινή κατάσταση. Έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ θαραλέο λαό, ο οποίος αντιδρά. Όλοι μας από όλες τις πλευρές της κοινωνίας συνεργαζόμαστε στους δρόμους, στις διαδηλώσεις αυτές και ελπίζουμε στη δική σας προσβλέπουμε στη δική σας πολιτική βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον κύριο Γκάλιον, τον κύριο καθηγητή να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Μικρόφωνο παρακαλώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας καλέσατε να μιλήσουμε ενώπιόν σας για έναν αγώνα που όλοι βλέπουν πόσο σήμερα είναι ιερός. Ο αγώνας μιας χώρας για τη μετάβαση, μιας χώρας που υπέφερε τόσο πολύ από ένα ε, μη δημοκρατικό και αυθαίρετο καθεστώς προς μια δημοκρατία, από μια δικτατορία προς μια δημοκρατία. Η Συρία, όπως οι πάντες γνωρίζουν, είναι μια χώρα ε, χίλιετιών που ανέκαθεν ε, είχε τον τρόπο να συμπεριλαμβάνει, να εντάσσει στην κοινωνία της όλες τις κοινότητες και να τις κάνει λαό, έθνος, ε, με σήμα το πνεύμα ε, της ανεκτικότητας, ειρήνης και μεγάλο ήθος πολιτών. Έπεσε θύμα ενός σοβιετικού τύπου καθεστώτος. Το κόμμα Μπαθ εγκαθίδρυσε ένα καθεστώς με καταστολή όλων των ελευθεριών, όλα τα δικαιώματα ε, παραβιάζονται και καπατούνται ακόμα και σήμερα και ο κόσμος ε, ε, ταπεινώνεται συστηματικά. Δυστυχώς η ευρωπαϊκή πολιτική τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια δεν ήταν άσχετη προς την κατάσταση αυτή η διατήρηση και η ιδέα της διατήρησης της σταθερότητας πάση θυσία και με κάθε τίμημα σε μια περιοχή όπου βρίσκονται τα δύο τρίτα των αποθεμάτων υδρογονανθράκων και όπου πάντα αυτό που προείχε ήταν η ασφάλεια του Ισραήλ συνεισέφεραν πραγματικά αυτοί οι παράγοντες και οφείλουμε να το θυμίζουμε αυτό. Ελπίζω σήμερα να ληφθεί κάποια απόφαση να τερματιστεί η πολιτική αυτή που ευνόησε ένα σύστημα δικτατορικό. Ο Άσαντ και ε, το καθεστώς του ανέκαθεν θεωρεί το πυλώνα σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Σήμερα είναι η πηγή όλων των ταραχών και όλες τις αστάθειες που ζουν οι Σύριοι, αλλά όχι μόνο και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης που ο Συριακός λαός δεν ε, είχε ποτέ τόσο στένος, δεν ήταν ποτέ τόσο αποφασισμένος να αποσπάσει τα δικαιώματά του δεν ήταν ποτέ τόσο έτοιμος να κάνει όλες τις θυσίε που χρειάζονται για να καθορίσει το μέλλον του και να ξεφορτωθεί το καθεστώς αυτό. Και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι ουδέποτε ένα καθεστώς δεν έδειξε τόσο μεγάλη βαρβαρότητα απέναντι στις προσδοκίες ενός λαού όπως αυτό δεν είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε. Ξέρουμε, πιστεύουμε ότι έχετε πολλή ενημέρωση για το τι συμβαίνει στη Συρία, αλλά για να σας ζητήσουμε να ε, δώσετε την υποστήριξή σας στην επιλογή του λαού αυτού. Να έχει το καθεστώς που του αξίζει. Δηλαδή, ένα καθεστώς που να απαντά στην επιλογή του λαού να εκπροσωπείται από μια εκλεγμένη κυβέρνηση από το λαό, που να εκπροσωπεί το λαό. Η Συριακή αντιπολίτευση χρειάστηκε χρόνο για να οργανωθεί. Σήμερα οργανώνεται. Γίνονται και έχουν ήδη γίνει πολλές ε, διασκέψεις για να ξεκαθαριστούν οι θέσεις και να καθοριστούν τα ρεύματα και σήμερα και αύριο ε, θα ακολουθήσουν και άλλες συσκέψεις, αλλά η Συριακή Αντιπολίτευση δεν είναι ουσιαστικά διχασμένη όπως συχνά ακούμε. Είναι απλώς πολυσχηδής και είναι φυσικό. Κάθε αντιπολίτευση είναι πολυσχηδής. Η ενωμένη αντιπολίτευση είναι μάλλον ενωμένη σε μια πλατφόρμα, σε μια βάση που μπορούμε να τη συνοψίσουμε ως εξής. Πρώτον, το σύνολο της αντιπολίτευσης συμφωνεί για μια μετάβαση προς ένα δημοκρατικό καθεστώς. Δηλαδή, σύσσωμη η αντιπολίτευση σήμερα απορρίπτει οποιοδήποτε συμβιβασμό με το σημερινό καθεστώς. Δεύτερον, σύσσωμη η αντιπολίτευση απορρίπτει κάθε είδους στρατιωτικής επέμβασης έξωθεν. Οι Σύροι, όλοι οι Σύροι συμφωνούν στην απόρριψη αυτής της εξωτερικής στρατιωτικής επέμβασης. Είναι βέβαιο ότι μπορούν με τα ίδια τους τα μέσα και τις δυνάμεις τους να φέρουν εις πέρας ε, αυτή την προσπάθεια και να τερματιστεί αυτό το δικτατορικό καθεστώς. Τρίτον, όλοι οι Σύροι συμφωνούν και θεωρούν τη Συρία ένα ενιαίο ενωμένο έθνος, ένα ενιαίο κράτος και μια ενιαία χώρα και απορρίπτουν κάθε είδους διάκριση ε, εθνοτική, ε, θρησκευτική ή οποιαδήποτε άλλη. Απορρίπτουν κάθε είδος διάκρισης και κάθε είδους κινητοποίησης ή υποδάβλησης τέτοιων αισθημάτων ή τέτοιων συμπεριφορών που προσπαθεί με κάθε τρόπο να τονίζει το καθεστώς ε, για να αντιμετωπίσει την ε, αύξηση της δύναμης της αντιπολίτευσης. Τέταρτον, σύσσωμη η αντιπολίτευση συμφωνεί και υποστηρίζει την ιδέα ότι οι διαδηλώσεις και η ε, αντιπολίτευση θα πρέπει να είναι πάντα ειρηνική στη συμπεριφορά της κάθε διαδήλωση, κάθε εκδήλωση και εκεί μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά είναι ενωμένη η αντιπολίτευση. Τώρα, τι ζητάει ο Συριακός λαός και η Συριακή αντιπολίτευση από τους Ευρωπαίους. Νομίζω ότι το βασικό είναι να κοιτάξουμε μαζί σας ποια μέτρα μπορούμε να βρούμε για να βοηθήσουμε το Συριακό λαό να υλοποιήσει τις ε, φιλοδοξίες και τις προσδοκίες του για τη μετάβαση προς ένα δημοκρατικό καθεστώς. Παράδειγμα, ακόμα και η παρουσία πολιτικών βουλευτών επιτόπου θα μπορούσε να είναι πολύτιμη για την προστασία των διαδηλωτών και παρακαλώ τα πολιτικά κόμματα να σκεφτούν νέες πρωτοβουλίες. Αλλά συνολικά η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να βοηθήσουν να σκεφτούν για τη δημιουργία κάποιων υπηρεσιών που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις ή απαντήσεις πρακτικής φύσεως, όσο και γρήγορες, στις επιτακτικές ανάγκες των ε, σύρων σε αυτή τη πολύ δύσκολη μεταβατική περίοδο. Σε εσάς εναπόκειται να ε, δείτε, να εξετάσετε με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε το λαό ε, για να βγει από αυτή τη φάση τόσο δύσκολη που διανύει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μάριο Νταβίτ, που όπως είπα είναι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον δόκτωρα Αλμαλέ και τον καθηγητή Γκαλιούν για τις ε, παρουσιάσεις τους, για τις μαρτυρίες που κατέθεσαν και θα ήθελα να εκφράσω τη γνώμη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή και παρακολουθεί εξαιρετικά προσεκτικά όλα τα γεγονότα στη Συρία και θα στηρίξουμε οποιοδήποτε κίνημα, οποιοδήποτε διάβημα που θα βοηθήσει να σταματήσει αυτή η δολοφονική αιματοχυσία στη Συρία και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο έδαφο, να διαμορφώσουμε τι προποθέσει για την εγκαθίδρυση τη δημοκρατία. Γιατί, όπω είπατε, έχουμε πολλέ κοινέ αξίε. Θα ήθελα να υποβάλω δύο-τρει ερωτήσει. Κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε σε συγκεκριμένα μέτρα ή σε συγκεκριμένα διαβήματα που θα μπορούσαμε εμείς και όταν λέω εμείς δεν εννοώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα μπορούσαν να αναλάβουν και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμβάλλει αλλά κάποια συγκεκριμένα μέτρα, κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο, την Επιτροπή να προβούν σε διαβήματα προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους ε, να σταματήσει η αιματοχυσία να εξασφαλιστεί η ειρηνική μετάβαση σε μια πιο ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία και κράτος γιατί ε, περισσότερη δημοκρατία δεν έχει νόημα δεν μπορούμε να έχουμε όλη δημοκρατία είναι δημοκρατική μια κοινωνία και μια χώρα ή δεν είναι υπάρχουν ε, κάποιες ενδείξεις ε, από τις Ιρανικές αρχές ε, ως προς αντιδράσεις της Συρίας υπάρχει κάποια θέση της Ιρανικής ε, κυβέρνησης ό,τι αφορά την καταστολή που επιβάλλει η Συρία στο λαό της σε ό,τι αφορά ε, το αίτημα για ειδικά μέτρα από το δικαστήριο του Λιβάνου υπάρχει κάποιος κανόνας, κάποια απόφαση για το ρόλο που διαδραματίζουν οι Συριακές Αρχές σε αυτό το θέμα. Και τέλος, μερικές φορές για να αποσπαστεί η προσοχή του κοινού από, μια κατάσταση, την κατάσταση στη χώρα μπορεί να γίνουν διάφορες κινήσεις ε, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Ισραήλ. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Ο κύριος Πέτερινγκ τώρα, που είναι πρόεδρος ομάδας εργασίας για τη Μέση Ανατολή. Παρακαλώ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μεγάλη εντύπωση μου προκάλεσαν τα όσα άκουσα από τους δύο καλεσμένους μας και θα ήθελα προσωπικά να σας πω ότι είμαι στο πλευρό σας ε, παραστάτης ε, με πλήρη αλληλεγγύη. Αναφερθήκατε στη σταθερότητα. Σταθερότητα ανήκει και ελευθερία και δημοκρατία τη δεκαετία του 70 στην Ευρώπη όταν υπήρχε ο κομμουνισμός πάντα και τότε μιλούσαμε για σταθερότητα. Αλλά ήταν μια σταθερότητα ησυχία κημητηρίου. Γι' αυτό σας ευχόμαστε η δημοκρατία να πετύχει. Και όταν μας λέτε τι μπορούμε να κάνουμε, ε, θέλουμε να κάνουμε κάτι αλλά χωρίς πίεση ε, χωρί βεβαιασμένε κινήσεις. Δεν θέλουμε να αναμειχθούμε, αλλά να σας βοηθήσουμε όταν εσείς μα ζητήσετε συγκεκριμένη βοήθεια. Έχω λοιπόν εδώ μια ερώτηση και θα ήθελα σύντομα να σας αναφέρω το εξή. Το έτος 2008, που ήταν το έτος του διαλόγου των πολιτισμών, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήρθε ε, και μίλησε ο Χασούν, ο μέγας μουφτής της Δαμασκού. Ήταν θαυμάσια ομιλία, συνεργασία των περιφερειών, των ε, πολιτισμών κτλ. Πριν από λίγες εβδομάδες σας απίφθηνα, μία, ε, απίφθηνα σε εκείνον μία επιστολή και του είπα να έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους των χριστιανικών εκκλησιών και να ζητήσει, να καλέσει να σταματήσει βία. Και μου απάντησε υπερασπιζόμενος το καθεστώς. Και ρωτώ, ε, οι διάφορες Ισλαμικές ομάδες εκεί πώς είναι. Ξέρουμε ο πρόεδρος Ασάτ ε, ε, και ο δικτάτορ με τους Αλεβίτες υπερασπίζονται την εξουσία τους. Αλλά τι γίνεται με τους Σουνίτες που είναι η μεγάλη πλειονότητα. Η δημοκρατική τους αίσθηση ποια είναι. Και τι γίνονται οι χριστιανοί. Είναι πολύ μεγάλη ανοχή για τους χριστιανούς στη Συρία. Πολύ με εξέπληξε αυτό. Και σε μια εκκλησία στη Δαμασκό υπάρχει σταυρός που φωτίζεται. Σε πολλές άλλες αραβικές χώρες αυτό δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, ε, οι ηγέτες, οι θρησκευτικοί, οι επίσκοποι των θρησκευτικών ε, κοινοτήτων εκεί των χριστιανών, πώς συμπεριφέρονται. Και δεν μιλώ μόνο για, την για το μυαλό αλλά και για την καρδιά. Πραγματικά είμαστε στο πλευρό σας ε, και συναισθηματικά ε, και με τη λογική και θέλουμε να γίνει δημοκρατία. Ο κύριος Μπέλντερ, ο οποίος είναι συντονιστής ε, τίνος, της ομάδας του και πρόεδρος της αντιπροσωπείας με το Ισραήλ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς τους εξέχοντες σύρους προσκεκλημένους μας. Και έχει σχέση με αυτό που είπε ε, ο κύριος Πέτερινγκ με τόσο ωραίο τρόπο. Εγώ έχω ένα πολύ καλό φίλο αραβιστή που μιλάει στα αραβικά. Είναι επιστήμονας, ζει εδώ και χρόνια στη Δαμασκό και ανησυχεί πάρα πολύ για την κατάσταση των εκκλησιών και των χριστιανών σήμερα στη Συρία. Και σας ρωτώ για την πολίτευση τι λέει, γιατί είναι βαθιά η αγωνία. ακούμε ε, για διάφορες βιαοπραγίες, ε, για τα επεισόδια και μας προβληματίζει πάρα πολύ. Πρόσφατα, χτες μάλιστα, έλαβα ένα έγγραφο από ε, χριστιανούς, οπαδούς εκκλησιών που μας δίνουν παραδείγματα τα οποία τονίζουν τους φόβους και την αγωνία. Με διάφορα συνθήματα για το τι θα πάθουν οι χριστιανοί όταν φύγει ο Ασάντ. Εσείς τι λέτε, πώς θα προστατεύετε. Η Συρία ξέρουμε ότι είναι μια περίπλοκη χώρα με πολλές θρησκείες, με πολλές εθνότητες. Τι σκέφτεστε για τη θέση της κουρδικής μειονότητας. Αυτό δεν είναι ευκαταφρόνητο. Και ε, είπατε και κάτι για την έξωθεν επέμβαση. Θέλετε να την αποφύγετε. Αλλά η κατάσταση είναι τέτοια ε, ώστε υπάρχει ήδη επέμβαση από εξωτερικούς σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συγκεκριμένα δεν επεμβαίνει, δεν έχετε εσείς Και επίσης τι γίνεται με τους εξτρεμιστές, τους τζιχαδιστές που ε, υποδαβλίζουν αυτά τα επεισόδια και ποντάρουν στην κλιμάκωση της κατάστασης στη Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φλότ που είναι πρόεδρος, πρόεδρος της ε, Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Τουρκία. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που ήρθατε στη συνεδρίαση. Φαντάζομαι λάβατε γνώση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Συρία και θα διαπιστώσατε πόσο στηρίζουμε με πυγμή και στένος στα κινήματα υπέρ της ελευθερίας και καταδικάζουμε απερίφραστα τη χρήση βίας, αλλά όπως είπατε κι εσείς δεν υπήρχε καμία έκκληση προς τον Μπασάρα Λασάντ να εγκαταλείψει τη θέση του, να εγκαταλείψει την εξουσία, ούτε αναφέρθηκε το υποτιθέμενο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας όπως τεκμηριώθηκε από τη Human Rights Watch ότι αφορά τη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων από το καθεστώς και οι ερωτήσεις των συναδέλφων δείχνουν ακριβώς τα όρια της υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί όλοι προβληματιζόμαστε για το τι μέλη μετά ε, και μας εξηγήσατε καταρχήν για το διάλογο. Είπατε ότι ίσως υπάρχει υπάρξουν κάποιε αντίφασει. Γιατί αν λέμε ότι ο πολιτικό διάλογο υπόκειται σε μια σειρά όρων, αυτό μα είπατε κύριε Αλμαλέχ, αποφυλάκηση των διαδηλωτών, απομάκρυνση των τάξ, κατάπαυση των βιοπραγιών. Αυτό δείχνει διάθεση διαλόγου. Ε, σε περίπτωση που εκπληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις υπάρχει δυνατότητα διαλόγου με το καθεστώς. Αλλά είπατε ότι είναι αδύνατος. οποιοδήποτε διάλογος με το καθεστώς δεν είναι αντίφαση, κάτι τέτοιο. Γιατί η κατάσταση δεν είναι διόλου απλή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μας διευκρινίσετε τη θέση σας. Στη Δαμασκό δεν έγιναν κάποιες απόπειρες διαλόγου και αν ναι, με ποιο κόμμα. Επίσης, μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω από το καθεστώς. Για παράδειγμα, στο στρατό ή σε άλλα σώματα που πρόσκειται στο καθεστώς υπάρχουν ε, αντίθετες φωνές, υπάρχουν κάποιες τριβές, υπάρχουν κάποιες λιποταξίες μιλήσαμε για τους ελεύθερους σκοπευτές του Ιράν, του Σνάιμερ. Τα καταλάβαμε αυτά, αλλά τι είδου συμμαχίες μπορούμε στο μέλλον να, να δημιουργηθούν σε περιφερειακό επίπεδο μετά από ανατροπή του καθεστώτος και ποιες θα είναι ίσως οι επιπτώσεις στην σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στην Αγγής Ανατολή. Ε, πώς θα μπορέσουμε επιχειρησιακά να ενισχύσουμε την ε, υποστήριξή μας ε, προκειμένου να εγκριθεί και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ένα ψήφισμα για τη Συρία για να διευκρινιστεί η απερίφραστη υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας με ένα αίτημα αποχώρησης του Μπασάρα Λασάντ από την εξουσία. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία άσκησε ισχυρότητε πιέσεις και επανειλημμένως υπέβαλε εκκλήσεις και μάλιστα σκεφτήκαμε ότι θα υπήρξε κάποιες προτάσεις εκδημοκρατισμού του καθεστώτος και βέβαια παρόλα αυτά έγινε και μια προσπάθεια για να διοργανωθεί και μια συνεδρίαση. Προσπαθεί η Τουρκία να δώσει με ένα νέο χαρακτήρα στις σχέσεις, γιατί είχε με το παλιό καθεστώς πολύ στενές σχέσεις και τώρα προσπαθεί να επαναπροσδιοριστεί κατά κάποιο τρόπο η Τουρκία. Τι περιμένετε εσείς από ένα τόσο ισχυρό και σημαντικό γείτονα όπως η Τουρκία που ούτως ή άλλως έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη ζώνη και περιοχή. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο και ένα δεκάλεπτο και στους δύο προσκεκλημένους για να απαντήσουν. Διαπιστώνεται ότι είναι ζωηρότατο το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το αποδεικνύουν οι ερωτήσεις που τέθηκαν. Ο δόκτωρ Αλμαλέχ και μετά ο καθηγητής Γκαλιούν. Πολλά ελέγχθησαν για τις διάφορες εθνότητες ή εθνοτικές μειονότητες, για τους χριστιανούς, για τους κούρτους. και θα ήθελα να πω ότι δεν υφίσταται πρόβλημα ως προς αυτό το σκέλος. Πριν από ε, μερικές ημέρες διάβασα τα απομνημονεύματα μετά του ε, Μαρούφ Αλ-Λιολίμπη. Όπως ξέρετε, διετέλεσε Πρωθυπουργό πολλές φορές στη Συρία. Μίλησε για τις, διαπρα... Ε, διαπραγματεύσεις με τους Γάλλους το 1936. Έκτοτε, πολύ εκτός Συρίας, πολύ συγγραφής, είχαν ζητήσει από τις γαλλικές αρχές να μην εγκαταλείψουν τη Συρία γιατί διαφορετικά οι χριστιανοί και άλλες θρησκευτικές εθνότητες θα διατρέχουν κίνδυνο. Αυτό ήταν μια μεγάλη, ένα μεγάλο ψέμα. Τώρα το καθεστώς παίζει το ίδιο παιχνίδι καλωσορίζω τα πολιτικά πρόσωπα και τις εφημερίδες των τύπου στα γραφεία μου εδώ και 15 χρόνια. Πάντα ακούω την ίδια εποδό. Τι θα κάνετε για τους χριστιανούς. Θα ήθελα να σας πω ότι στις απαρχές της δημοκρατίας της Συρίας ο πρωθυπουργός, ο Φάρσελ Χούρι, ήταν χριστιανός. Κανένας δεν είπε γιατί ο Φάρσελ Χούρι ήταν πρωθυπουργό. Ο Γάσαν Μελετάση ήταν πρόεδρος, ο οποίος αποχώρησε. Ο Φάρσελ Χούρι έγινε πρόεδρος της Συρίας, ο οποίος ήταν χριστιανός. Δεν συνέβη τίποτα. Κανένας δεν προέβαλε αντίρρηση για λόγους θρησκευτικούς, εθνοτικούς και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια ειρηνική συμβίωση στη Συρία. Το καθεστώς του Ασάντ, ειδικά το καθεστώς του Ασάντ δημιούργησε αυτό το προηγούμενο ότι είμαστε κατά των, ε, των, των χριστιανών ή των μουσουλμάνων. Εμείς στην αντιπολίτευση συνεργαζόμαστε με τους πάντες. Έχουμε και δρούζους, έχουμε και χριστιανούς. Τι σημαίνει αυτό. Όλοι είμαστε Σύριοι. Και στη, στην επανάσταση όλοι λέμε «wahed», δηλαδή ότι όλη η Συρία είναι μία, ενιαία. Αυτό μπορώ να σας πω και δεν χρειάζεται επεξηγήσεις. Δεν θεωρούμε ότι πρόκειται για κάποιον κίνδυνο. Ο δάσκαλός μου ήταν ο Μουστάφα Σιβάη ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της μουσουλμανικής αδελφότητας. Ήταν μέλος του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, το μεταξύ 1945 και 49 μετά το πραξικόπημα, δηλαδή μέχρι να γίνει το πραξικόπημα το 49, ο δάσκαλός μου της μουσουλμανικής αδελφότητας ήταν στο κοινοβούλιο, ήταν βουλευτής. Αυτά δεν τα σκεφτόμαστε, δεν τα συζητάμε. Όμως ήταν πραγματικότητα. Πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι θετικό για όλους τους πολίτες. Διότι διαβιούν υπό άσχημες συνθήκες όλοι, ανεξαιρέτως. Θεωρούμε όλοι ότι είμαστε εργαζόμενοι στην γεωργική εκμετάλλευση του Ασάντ. Δεν δεχόμαστε αυτό τον τρόπο ζωής. Όλοι οι Σύριοι, όλοι οι πολίτες, από όπου και αν προέρχονται, θέλουν να αλλάξουν την ποιότητα ζωής τους, να έχουν ελευθερία, να μπορούν να εκφραστούν ανεξάρτητα από το που προέρχονται. Και άρα δεν τρέφουμε κανέναν φόβο από αυτή την πλευρά. Μερικοί φίλοι μίλησαν για το Ιράν δηλαδή πώς δρά και πώς συμπεριφέρεται έναντι της Συρίας. Κατά την άποψή μου και πολλά μέλη επίσης της αντιπολίτευσης πιστεύουν ότι το Ιρανικό καθεστώς βοήθησε το δικό μας δικτατορικό καθεστώς διότι και τα δύο καθεστώτα έχουν το ίδιο υπόβαθρο. Είναι δικτατορικά καθεστώτα. δηλαδή το παρελθόν ήταν του, το παρελθόν του Αγιατολάχ. Είναι δικτατορικό καθεστώς. Ήταν και είναι. Και το ίδιο ισχύει και για την οικογένεια Ασάντ, η οποία έκανε αυτή την, ε, αυτό, έδωσε αυτό το αλληλένδετο στοιχείο, έτσι ώστε να μπορούν να προσέρχονται οι Ιρανοί και να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί είναι και τα δύο δικτατορικά καθεστώτα πολλά επαναστατικά στοιχεία προσήλθαν από το Ιράν για να βοηθήσουν το δικό μας καθεστώς. Μιλώ για το, τη θρησκευτική επανάσταση, τους φρουρούς της επανάστασης. Και, και δύο μέλη από την Χεσμολά από το Λίβανο επίσης προσήλθαν για να βοηθήσουν το δικτατορικό μας καθεστώς διότι προασπίζουν τα δικά τους συμφέροντα. Η Συρία αποτελεί την ε, γεφύρωση μεταξύ του Ιράν και της Χέσμπολα στο Λίβανο. Γι' αυτό θέλουν τη διαιώνιση αυτού του καθεστώτος. Εμείς όχι. Εμείς το άκρο αντίθετο. Εσείς μας μιλήσατε για τις διαπραγματεύσεις, το διάλογο με το καθεστώς. Το καθεστώς προσκάλεσε ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης, αλλά κανένας δεν δέχτηκε αυτό το διάλογο με ένα καθεστώς που φωνεύει. Εδώ και τρεις μήνες ζητήσαμε από το καθεστώς ότι αν θέλει να προωθήσει το διάλογο, θα πρέπει να απομακρυνθούν τα τάγκς, οι ένοπλες δυνάμεις. Οι μυστικές δυνάμεις δεν πρέπει να βασανίζουν τους ανθρώπους. Να μπορούν οι άνθρωποι να διαδηλώνουν ειρηνικά. Να ελευθερώσουν τους φυλακισμένους. Τώρα έχουμε 15.000 φυλακισμένους. Και στο παρελθόν είχαμε 5.000 Δηλαδή μιλάμε για 20.000 πολιτικούς κρατουμένους. Εξαιτίας των πεπιθήσεών τους δηλαδή φυλακίζονται χωρίς κατηγορίες. Όμως το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται για την ένομη τάξη, για την εφαρμογή του νόμου. Εμείς από πλευράς αντιπολίτευσης θέλουμε να δούμε ποια είναι η θέση των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, υπάρχει η μία πτέρυγα που απαρτίζεται από 60.000 που προστατεύουν το καθεστώς τον Πρωθυπουργό. Πρόκειται για 60.000 που βρίσκονται πολύ κοντά στην οικογένεια Ασάντ. Θα συνεχίσουν με αυτή τη στάση, αλλά το ίδιο δεν ισχύει για την άλλη πτέρυγα των ενόπλων δυνάμεων. Γι' αυτό και βλέπετε πολλούς στρατιωτικούς που εγκατέλειψαν εγκατέλειψαν ε, τις ενοπλές δυνάμεις και θα μεταβούν και στην Τουρκία. Μετέβησαν στην Τουρκία και θα τους συναντήσω σε λίγες ημέρες. Και νομίζω ότι ο στρατός θα σταματήσει κάποια στιγμή το καθεστώς δεν θα επιτρέψει πλέον την ε, αιματοχυσία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ θετικό αυτό το τελευταίο που είπατε, γιατί σε όλες τις κοινωνίες ο στρατός είναι ο ισχυρότερος κλάδος. Παρακαλώ, ο καθηγητής Γκαλιού. Ε, Euh, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίπλοκη και βεβαίως υπάρχουν και τάσεις διαθρησκευτικές, θα το συζητήσουμε και αυτό. Νομίζω τέσσερα ή πέντε είναι τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις. Το θέμα των μειονοτήτων και των, της πλειοψηφίας της πλειονότητας, κάποιος το έθεσε βεβαίως, γιατί μετά σαν εποχή είναι σημαντικό. Το δεύτερο, εξωτερική επέμβαση και αν υπάρχει εξωτερική επέμβαση παρέμβαση ιασδήποτε μορφής. Το τρίτο, διάλογος με την εξουσία, πώς το βλέπει η αντιπολίτευση και πώς σήμερα θεωρεί τη σχέση της με το καθεστώς. Τέταρτον, ε, λίγο για τις ένοπλες δυνάμεις στο στρατό, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάποια στοιχεία. Και το πέμπτο είναι οι μελλοντικέ συμμαχίες. Και είναι σημαντικό εξωτερική πολιτική και η θέση των περιφερειακών δυνάμεων και ο ρόλος της Τουρκίας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Λοιπόν, για το θέμα ε, της πλειονότητας και των μειονοτήτων. Νομίζω ότι υπάρχει ένα στοιχείο ιστορίας εδώ. Η Συρία δεν γνώρισε ποτέ θρησκευτικές διαμάχες. Είναι η μόνη χώρα ουδέποτε ε, στην ιστορία της. Είναι σταυροδρόμι πολιτισμών και η ίδια της η ταυτότητα βασίζεται σε αυτό ε, το είδος της πολυφωνίας, τον πλουραλισμό. Και είναι και θέμα αγωγής του πολίτου. Μαθαίνουν οι πολίτες να συμβιώνουν, να συνδιαλέγονται ε, και είναι η μόνη χώρα που δεν έχει ένα ηγέτη της ανεξαρτησίας της, αλλά τέσσερις. Και ο σημαντικότερος ε, προέρχεται από την πιο ε, μικρή μειονότητα, Δρούζος, ο αρχηγός της Επανάστασης της Ανεξαρτησίας, με έναν Κούρδο με ένα Λεβίτη και με ένα Σουνίτη. Τέσσερις είναι οι ηγέτες της ε, ανεξαρτησίας και ποτέ κανένας από τους τέσσερις δεν θεώρησε τον εαυτό του ε, μέλος κάποιας μειονότητας, παρά μόνο Σύρο. Και η εθνική γιορτή εορτάζεται από όλους. Από αυτή την τετραμελή ηγεσία ε, είναι η μόνη χώρα την περιοχή που είχε μετά την ανεξαρτησία τον πρώτο πρωθυπουργό χριστιανό, τον Φαρές Αλχούρη. Αυτά είναι στοιχεία που δείχνουν κάπως τη γενική ατμόσφαιρα και το κλίμα το πολιτισμικό στο οποίο ε, διαβιούν οι Σύροι. Δεν υπάρχουν εμπόδια και φραγμοί μεταξύ των Σύρων ανάλογα με τη θρησκευτική ταυτότητα του καθενό. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, κοινωνιολογικό αν θέλετε επιχείρημα, στη Συρία δεν υπάρχει ελίτ που να ε, είναι χωρισμένη σε φυλές, σε ομάδες, κλάν, γιατί εκεί είναι ε, το επικίνδυνο. Οι Αλεβίτες όταν έχουν ε, μια πολιτική ελίτ, το ίδιο οι Σουνίτες, το ίδιο οι Χριστιανοί. Δεν υπάρχει τέτοια κάθετη ελίτ. Ανέκαθεν η ελίτ στη Συρία ήταν ενωμένη και σήμερα ενωμένη στο ίδιο κόμμα. Δεν υπάρχουν ε, θρησκευτικά κόμματα. Εκτός από το κουρδικό κόμμα που εκπροσωπεί μια ε, εθνική μάλλον ευαισθησία και όχι εθνοτική. Άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, στην ιστορία μας και στην κοινωνιολογία της Συρίας νομίζω είναι πολύ μικρός ο κίνδυνος να υπάρξουν θρησκευτικές ε, συγκρούσεις ή και πόλεμος. Μπορεί λόγω της σημερινής κατάστασης να παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Βεβαίως και οι Αλεβίτες ανησυχούν και οι Χριστιανοί έχουν ε, ανατραπεί τα πράγματα ε, ε, το καθεστώς τους έχει βάλει στο μυαλό ότι εκείνο τους προστατεύει, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας δεν τους προστάτευαν οι μουσουλμάνοι γιατί δεν αυτό προσδιορίζονταν ως φίλο μουσουλμάνοι ή αντιμουσουλμάνοι, αλλά τους προστάτευε ο ρόλος που διαδραμάτιζαν στην πολιτική ζωή του τόπου, στην απελευθέρωση του τόπου, στην οικοδόμηση του τόπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και έτσι βλέπει η ελίτ τα πράγματα ακόμα και σήμερα. Και αυτό είναι εγγύηση απέναντι σε κάθε διχασμό. Καλά, σήμερα μπορεί να έχουμε μικροεπισόδια μεμονωμένα, Ε, αν αυτά παρατηρηθούν θα επέμβει η ελίτ και η χριστιανική και η μουσουλμανική κλπ. Στη Λατάκια τι έγινε. Προσπάθησε το καθεστώς να σπείρει ε, ζυζάνια και συναντήθηκαν οι ουλεμάδες και των δύο κοινοτήτων για να ε, σημάνουν συναγερμό και αποφάσισαν ότι κάθε ημάμις, κάθε κοινότητα θα διευθύνει την προσευχή ε, στα τεμένη της άλλης κοινότητας και έτσι αποσοβήθηκε αυτός ο κίνδυνος. Είναι πραγματικά θησαυρό η ευφυΐα που έχουν σε αυτά τα θέματα οι Σύροι και δεν θα πέσουμε σε θρησκευτική σύραξη, σας διαβεβαιώ. Οι μουσουλμάνοι βεβαίως σήμερα όπως και σε πολλές άλλες, ίσως όλες αραβικές χώρες, έχουν ε, ε, κάποια θρησκευτική ευαισθησία και στην Τουρκία και σε δημοκρατικές χώρες θα έλεγα. Αλλά από τότε που εμφανίστηκε το κόμμα του Ερντογάν στην εξουσία δεν κυριαρχεί πλέον το ιρανικό μοντέλο στο μυαλό των ε, μουσουλμάνων και των Ισλαμιστών συμπεριλαμβανομένων. Έχουν στο μυαλό τους το τουρκικό μοντέλο. Ανακάλυψαν οι μουσουλμάνοι απανταχού της γης ότι υπάρχει ένα μοντέλο το τουρκικό που συμφιλιώνει το Ισλάμ με τη δημοκρατία και λειτουργεί πολύ καλύτερα από ένα μοντέλο που μόνο συγκρούσεις έχει προκαλέσει εσωτερικές και εξωτερικές. Ψυχολογικά, πολιτικά και πολιτισμικά έχουν πάρει διαζύγιο το Ιρανικό μοντέλο. Παντού οι μουσουλμάνοι. Και δεν γίνεται λόγος για την Ισλαμική Επανάσταση, αλλά για μη, ε, θεοκρατικό κράτος, κοσμικό κράτος, ε, δημοκρατία κτλ. Και αυτό εμπνέει πολύ περισσότερο και τους λαούς και τις προσδοκίες, μεταξύ άλλων και τα Ισλαμιστικά κόμματα. ελπίζουν να ταυτιστούν με μία νέα τέτοια μορφή περισσότερο από ε, πολιτιστικά ή θρησκευτικά στοιχεία. Λοιπόν, ε, επόμενο θέμα. Η μετά Ασάντ εποχή. Ή μάλλον όχι, προηγουμένω οι έξωθεν παρεμβάσει υπάρχουν τέτοιε επεμβάσει. Εμεί νομίζουμε ότι οι Ιρανοί σίγουρα έχουν κάποια δράση και δεν το έκρυψε ο Σύρος Υπουργό Εξωτερικών. Το δηλώνει ο άνθρωπο ότι οι Ιρανοί μα βοηθούν. Τώρα πώ βοηθούν δεν ξέρω σίγουρα με συμβούλους ασφαλείας, με στρατιωτικούς συμβούλους, ενδεχομένως και κάποια άλλα στοιχεία. Δεν έχουμε ακόμα ακριβώς εντοπίσει Ιρανούς ως πρόσωπα που να δρούν επιτόπου και δεν νομίζω ότι μπορούμε να κατηγορούμε. Μπορεί ε, τα Υπουργεία Εξωτερικών των χωρών της Δύσης να γνωρίζουν περισσότερα, αλλά προς το παρόν είναι η ηθική υποστήριξη πολιτική και κάποια εμπειρογνωμοσύνη ε, και είναι και φυσιολογικό γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ε, σύμμαχο της, ε, του Συριακού καθεστώτος Ιρανή. Διάλογος λοιπόν με το καθεστώς τώρα. Μέχρι πρότινος οι Σύριοι πίστευαν όπως και οι Δυτικοί, ότι θα μπορούσαν να ποντάρουν στον Μπασάρ για να απεμπλακούμε λίγο από το παρελθόν, από την υπόλοιπη τάξη των προνομιούχων, των στρατιωτικών, ε, των μηχανισμών ασφαλείας, για να αρχίσει μια δημοκρατική μεταρρύθμιση. Απέτυχε. Και ο Μπασάρ απέτυχε. Δεν επέδειξε και καμιά τεράστια τη θέληση, ούτε δυνατότητα να απαγκιστρωθεί από τη στρατιωτικό ασφαλίτικη χούντα και να προχωρήσει προς τις προσδοκίες του λαού. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκφωνήσει λόγο στο λαό του. Στην αυλή του μιλάει και μόνο. Ποτέ δεν υποσχέθηκε δημοκρατική μετάβαση. Για μεταρρυθμίσεις μιλάει. Ούτε είπε ε, ποτέ ότι όταν ολοκληρωθεί η σημερινή μου θητεία που λύγει το 2014 γιατί έχει ακόμα μερικά χρόνια. Στο τέλος της θητεία μου θα αποχωρήσω από την εξουσία. Ουδέποτε δήλωσε ότι θέλει προεδρικές εκλογές με ε, αντιπάλους ε, και ένα ανταγωνισμό. Επίσης, συνεχίζει ταυτόχρονα να διατάσει να πυροβολούν τον πληθυσμό με πραγματικά πυρά. Σήμερα ε, είναι ακόμα πιο μεγάλη βία. Μπορεί να είναι λιγότερα τα πραγματικά πυρά, αλλά σαρώνουν ολόκληρες συνοικίες, σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα. Αυτό που είχε ε, υποσχεθεί ο Καντάφης στους Λίβιους, ότι θα σας βρούμε στα σπίτι, σπίτι, πόρτα-πόρτα, δρόμο-δρόμο, θα σας πιάσουμε, θα σας βασανίσουμε. Έχουν αρχίσει και σαρώνουν, ε, κόβουν το ρεύμα, το νερό, ε, το ίντερνετ, τα πάντα, για να απομονωθεί τελείως ο πληθυσμός και καταστολή, βίαιη. Ε, με βασανιστήρια. Μέχρι τώρα 53 νεκρούς είχαμε από βασανιστήρια στις φυλακές. 53 νεκρούς από την αρχή των γεγονότων. Για να μην μιλήσουμε για τις 15.000 φυλακισμένους και 2.000 μάρτυρες κτλ. Με ένα τέτοιο τύπο, ε, τι να πεις σήμερα αν οργανωμένη αντιπολίτευση δεχτεί το διάλογο ανεφόρων, γιατί αυτό θέλει το καθεστώ, αυτό μα ζητάει. Δηλαδή, θα εξακολουθήσω να σα πυροβολώ, να σαρώνω τι πόλει, να ε, ε συλλαμβάνω νέου, να του βασανίζω, αλλά ελάτε να μιλήσουμε. Ε, ποια πολιτική δύναμη αντιπολίτευσης μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο διάλογο χωρίς να χάσει ε, την αξιοπιστία της, το πρόσωπό της απέναντι στο λαό απλώς θα θεωρηθεί μια δύναμη που θέλει μερικές θεσούλες, καρέκλες. Αυτά τα τάζει ε, αβέρτα ο Μπασάρ. Μια Παρασκευή που ζητήσαμε να δια, ε, δηλώσει ο κόσμος, την ε, ονομάσαμε η Παρασκευή του μη διαλόγου. Δηλαδή δεν δεχόμαστε τέτοιες επιταγές για διάλογο, δεν είναι πρόσκληση αυτό, είναι ελάτε, αλλά εγώ θα σας πω ποιος θα είναι μέλος στην Επιτροπή ε, Προετοιμασίας του Διαλόγου. Θα γράψω την ημερήσια διάταξη, θα αποφασίσω ποια θα είναι αυτή και δεν ορίζει και το στόχο, το σκοπό. Γιατί να συζητήσουμε με πιο απότερο στόχο. Για να μοιράσουμε την πίτα ή να σκεφτούμε μια μεταβάση στη δημοκρατία. Όχι, εγώ θα αποφασίσω και ποιοι θα συμμετέχουν στο διάλογο. Δηλαδή η αντιπολίτευση αποκλείστηκε πλήρως και απολύτως από κάθε διάλογο, από κάθε συνεννόηση για να προετοιμαστεί αυτός ο διάλογος. Δεν δικτά διάλογος, είναι επιταγή, ε, που είναι χαρακτηριστική και για το καθεστώς αυτό. Είναι φυσιολογικό ο κόσμος δεν ε, απορρίπτει το διάλογο, Το ψευτοδιάλογο διάλογο ε, απορρίπτει, την παγίδα που στείνει στην αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε διάλογο χωρίς να σταματήσει πλήρως η καταστολή. Είναι εκ των όνων κάνεφα, διαπραγμάτευτο αυτό. Αν συνεχίσει η καταστολή, διάλογο δεν υφίσταται. Δεν μπορεί να ε, συνδιαλέγεσαι και να συνομιλεί ε, με το πιστόλι στον κρόταφο. Ε, αυτό είναι αυθαιρεσία και τίποτα άλλο. Λοιπόν, εδώ πιστεύω ότι η αντιπολίτευση συμφωνεί επ' αυτού και είναι ομόφωνη. Δεν συνομιλούμε με το καθεστώ. Γι' αυτό και ο διάλογο που οργάνωσε το καθεστώ ε, τη προάλλε απέτυχε παταγωδός καμία προσωπικότητα, κανένα μέλος, όχι μόνο των κομμάτων, δεν ομιλώ για τα κόμματα, καμία προσωπικότητα δεν εμφανίστηκε, ούτε δέχτηκε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο διάλογο. Έτσι, που να είναι γνωστή η προσωπικότητα τη αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι ήταν φιάσκο και το παραταγώδη αποτυχία του διαλόγου, διότι η προσφορά ήταν τελείω. Ε, χωρίς κανένα νόημα και κανένα ενδιαφέρον. Ο στρατός τώρα τι γίνεται, οι ένοπλες δυνάμεις. Ακούμε ότι περιμένει λέει ο λαό να δράσει ο στρατός κάποια στιγμή. Εγώ από την αντιπολίτευση δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπολογίζουμε στη διάλυση του στρατού. Όχι, θέλουμε ο στρατός να παραμείνει συμπαγής. Οι Σύροι δεν θέλουν να διαλυθεί ο στρατός. Είναι σημαντικός θεσμός για να ε, διαφυλάξει την τάξη μετά, στη μετά την Ασάντα εποχή. Ίσως και ο μόνος θεσμός. Και ο στρατός στο σύνολό του δεν συμμετέχει στην καταστολή. Είναι κάποιες μονάδες επίλεκτες παρακαλώ που τις στέλνουν ε, στα συγκεκριμένα σημεία. Και κάποια στιγμή ο Συριακός στρατός πιστεύω θα παίξει το ρόλο του. Πότε δεν ξέρω, αλλά θα παίξει το ρόλο του. Ίσως τώρα πρέπει να το πούμε. Ο Μπασάρ δεν έχει πια αξιοπιστία. Δεν μπορούμε να συζητούμε με τον Μπασάρ για να ηγηθεί ε, σε μια μεταβατική ε, ε, κατάσταση. Η μετάβαση νομίζω θα γίνει από ένα εθνικό συμβούλιο ή μεταβατικό όπου θα συμμετέχουν και οι ένοπλες δυνάμεις, οι στρατιωτικοί που δεν έχουν κάνει εγκλήματα βεβαίως και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης για να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας και να προετοιμάσουν την μετά Άσαντ εποχή στη Συρία. Στη δημοκρατία. Πέμπτο και τελευταίο λοιπόν, οι συμμαχίες. Νομίζω ότι μία από τις ιδιαιτερότητες της κρίσης στη Συρία είναι ότι οι περιφερειακές δυνάμεις υπολογίζουν πολύ στη Συρία, περισσότερο Μάλλον ε, μετράνε πάρα πολύ και η Τουρκία και το Ιράν και η Αίγυπτος παίζουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο για τη Συρία από ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και ε, η Ευρώπη. Και ζητώ συγγνώμη που τα λέω αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να συνεργαστούν με αυτές τις περιφερειακές δυνάμεις. Η μόνη λύση, κατά την άποψή μου, θα ήταν, γιατί είναι λάθος να γίνει το θέατρο των συγκρούσεων τώρα αυτών των περιφερειακών δυνάμεων η Συρία. Η λύση για τη Συρία περνάει μόνο μέσα από μία συνεννόηση, ένα διάλογο μεταξύ των περιφερειακών αυτών δυνάμεων. Και καλωσορίζω εγώ και χαιρετίζω την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ε, ο οποίος θα μεταβεί στο Ιράν, ο κύριος Νταβούτογλου, ε, και θα περάσει από τις χώρες του κόλπου και την Αίγυπτο. Νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξει ένα τέτοιο διάβημα. Συνεργασία των περιφερειακών δυνάμεων. Τουρκία, Ιράν και το θέμα αυτό να διαχωριστεί από τη διαφωνία που έχει το Ιράν με την Ευρώπη για τα πυρηνικά θα πρέπει να το κρατήσουμε ξεχωριστό. Για να λυθεί το ζήτημα της Συρίας, να βοηθηθεί η Συρία να βγει από το αδιέξοδο, θα πρέπει να συνεννοηθούν οι περιφερειακές δυνάμεις, να υπάρξει κάποια συνεννόηση, ένας διάλογος ε, ειδικά Ιράν και Τουρκίας και των χωρών του Περσικού κόλπου και της Αιγύπτου βέβαια, των Αράβων. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά πιστεύω ότι οι Ιρανοί δεν θα θεωρήσουν ότι η αλλαγή του συστήματος του καθεστώτος στη Συρία θα φέρει τη Συρία αντίπαλό τη. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ούτε αντίπαλος του Ιράν, ούτε κανενός άλλου κράτους. Θέλουμε σχέσεις συνεργασίας με όλες τις περιφερειακές δυνάμεις που να βασίζεται στο αμοιβαίο ε, συμφέρον, στον αμοιβαίο σεβασμό και νομίζω και εσείς μπορείτε να βοηθήσετε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Oh, Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Σε πολλές, είχα πολλές ευκαιρίες να συναντηθώ με τον ε, πρόεδρο ΣΑΤ και νόμιζα ότι, είχαμε, ότι είχε πολύ λιγότερη εξουσία από ό,τι νομίζαμε εμείς και νόμιζα ότι ήταν υπό την ε, κυδαιμονία του πατρός της παλιάς ε, φρουράς και ότι οι μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε τόσες πολλές φορές ε, δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν και νόμιζα ότι αυτό ήταν ο λόγος, λόγω της μικρής εξουσίας που είχε. Εν πάση περιπτώσει τώρα είναι πολύ αργά πια να μιλάμε γι' αυτό. Κάτι που δεν αναφέρθηκε εδώ είναι ότι όλοι ε, αποδοκιμάζουμε την υποκρισία της διεθνούς κοινότητας και το γεγονός ότι εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και νομίζω θα πρέπει να στυλιτεύουμε και να καταδικάζουμε τα μέρη της διεθνούς κοινότητας που ε, όπως η Ρωσία, η Βραζιλία ε, εκδηλώνουν τέτοια συμπεριφορά όταν μιλούμε για την ε, Συριανή κρίση και διαφορετικά την αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες από την κρίση στη Λιβύη. Τώρα, για το κοσμικό καθεστώς που είπαμε, κοσμικό κράτος ε, στη Συρία για το μέλλον. Νομίζω ότι ο διάλογος των πολιτισμών και ο διαθρησκευτικός διάλογος και η διαθρησκευτική συνύπαρξη μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων είναι κάτι που ε, αξιολογούμε πολύ θετικά στη Συρία και ελπίζω να συνεχιστεί. Τώρα, τηλεγραφικά, το θέμα των, της χθεσινής επίθεσης σε πρεσβείες. Φυσικά και αυτό το καταδικάζουμε δρυμύτατα και θα πρέπει να σκεφτούμε τι συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε ε, τι συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να σταματήσουμε την αιματοχυσία. Δεν νομίζω ότι με το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του Α ή του Β ή με τη τέτοια κατάσχεση μπορούμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Ούτε είμαι υπέρ της εισβολής στη Συρία ή με παρόμοια στρατηγική με αυτή που θετήσαμε στη Λιβύη. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει με πιο συγκεκριμένο τρόπο, πιο από τα μέτρα και να σας ζητήσω τέλος να μην χάσουμε τις επαφές μεταξύ μας και να σας ευχηθώ και προσωπικά αλλά ευχηθώ και στο λαό της Συρίας καλή επιτυχία στην μεταβατική αυτή περίοδο που διανύει η χώρα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκο, ευχαριστώ πολύ. Όπως διαπιστώνετε υπάρχει αλληλεγγύη από εμά και εκτιμούμε ιδιαίτερες πληροφορίες που μας δώσατε και μάλιστα το γεγονός ότι μας μεταφέρατε ένα κομμάτι της πραγματικότητας ε, στις γνώσεις που έχουμε για το τι συμβαίνει εκεί. Ήταν πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση και σας εύχομαι καλή επιτυχία.